Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη συνάντηση κορυφής λοιπόν. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να καλωσορίσω την εξοχότητά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη τιμή για μας να βρισκόμαστε για να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. που αφορά την οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων παραγόγων του άνθρακα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας. Ο ρόλος όλων σας, κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο, κύριε Πρόεδρε Φαν Ρομπέη, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσάς και όλους τους προσκεκλημένους μας σήμερα εδώ. Θα ήθελα να κάνω μια απλή δήλωση καταρχάς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πιο ευαίσθητη περιβαλλοντικά συνέλευση εκλεγμένων αντιπροσώπων στον κόσμο. Ήδη από τις πρώτες εκλογές μας άμεσες, άμεσης καθολικής ψηφοφορίας 1979 δημιουργήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ήταν η πρώτη φορά νομίζω στην κοινοβουλευτική ιστορία που οργανώσαμε μια τέτοια Επιτροπή έτσι ώστε να προωθήσουμε νομικές ρυθμίσεις. Αλλά για να υπάρξουν νομικές ρυθμίσεις απαιτούνται συναντήσεις, ανταλλαγές απόψεων εν μέσω των δημοκρατικών μας κοινωνιών και συναντήσεις όπως αυτή εδώ σήμερα. Οι ιδέες οι οποίες γεννιούνται σε τέτοιου είδους φόρα κατέστησαν τις νομικές ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος καλύτερες μέσω των συζητήσεών μας μπορούμε να καταλήξουμε σε λύσεις για τα προβλήματά μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ τον ε, συμπρόεδρο πρίγκιπα της Ουαλίας ο οποίος εμπλέκεται και στα θέματα του περιβάλλοντος και στα θέματα των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών εδώ και 25 χρόνια και στην καθημερινότητά του και μέσω των φιλανθρωπικών οργανώσεων στις οποίες εμπλέκεται η αυτού βασιλική εξοχότης δίνει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να ζήσει σεβόμενο στην φύση και να βοηθήσει να ζήσουν σωστά οι επόμενες γενιές. Να αναφερθώ σε μία μόνο από τις πρωτοβουλίες τους. Είναι το πρόγραμμα για την προστασία των τροφικών δασών του ε, του οποίου ηγείται. Εξοχότατε, ήσασταν εδώ πάλι μαζί μας εδώ και τρία χρόνια και είχατε πει στα μέλη μας ότι η ορολογιακή βόμβα της καταστροφής του ανθρώπινου κλίματος έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή να μας απειλεί. Λοιπόν, η νέα μας στρατηγική τώρα για την Ευρώπη του 2020 θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε με σωστές επενδύσεις στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες νέες καλύτερες συνθήκες. Αυτό το πρότεινε και στις 5 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελευταία και προσπαθούμε ακριβώς να σφραγίσουμε με την προσπάθειά μας αυτή όλες τις δραστηριότητες στην κοινή πολιτική στον τομέα της ενέργειας Κάτι τέτοιο δεν θα μας βοηθήσει μόνο να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, αλλά θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής ασφάλειας, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της ενέργειας, γιατί η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή την οποία δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και να παράγουμε. Και ακριβώς αυτή είναι η τριπλή στόχη που έχουμε για το 2020. Αυτή είναι στόχη περιβαλλοντική για όλο τον κόσμο άλλωστε. Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και 20% επίσης αύξηση ανανεώμενων ε, μορφών ενέργειας. Λοιπόν, θα πετύχουμε μια τέτοια οικονομία λοιπόν με χαμηλή απόδοση άνθρακα εφόσον υπάρξει σωστή συνεργασία ανάμεσα στους πολιτικούς και στις βιομηχανικές δραστηριότητες. Οι πολιτικοί θα πρέπει να δημιουργήσουν το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να λειτουργείται και ο επιχειρηματικός κόσμος θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ευαίσθητος περιβαλλοντικά και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας της βιομηχανίας είναι ανάμεσά μας σήμερα και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Οι ψηφοφόροι μας κυρίες και κύριοι είναι οι πελάτες σας και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι είναι οι ίδιοι αυτοί οι Ευρωπαίοι, τα εκατομμύρια Ευρωπαίοι που θέλουν να ζήσουν σε έναν κόσμο ο οποίος να είναι φιλικότερος περιβαλλοντικά. Εξοχότατε έχετε το λόγο.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 αερίων κατά 50% μέχρι το 2050. Αυτό σημαίνει ότι το 30% είναι μόνο ένας ελάχιστος στόχος. Κυρίες και κύριοι, ας μην ξεχάσουμε ότι η βιομηχανική γεωργία που εξαρτάται κατά πολύ από το πετρέλαιο και από την υψηλή απόδοση που τώρα κυριαρχεί στην παραγωγή τροφίμων στον κόσμο σχετίζεται με την τιμή του πετρελαίου. Μία μελέτη υπολογίζει ότι ένα άτομο με μία χαρακτηριστικά δυτική διατροφή καταναλώνει 4,4 λίτρα πετρελαίου την ημέρα και αυτός ο παράγων βοήθησε να αυξηθεί κατά πολύ ο δείκτης τροφίμων του Οργανισμού Διατροφής και Τροφίμων στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που δημιουργήθηκε το 1999. Θα πρέπει να ξέρουμε επίση ότι αυτό συμβαίνει ενώ ένα δισεκατομμύριο άτομα υποσυτίζονται και άλλο ένα δισεκατομμύριο πεινάει κάθε μέρα. Ενώ ένα άλλο δισεκατομμύριο υποφέρει από τις επιπτώσεις ε, της υπερδιατροφής και της παχυσαρκίας. Στις πλούσιες χώρες εκατομμύρια δολάρια τροφίμων σπαταλώνται και πετιούνται στα σκουπίδια κάθε χρόνο. Ενώ στον αναπτυσσόμενο κόσμο 40% των ε, γεωργικών προϊόντων πάνε χαμένα πριν φτάσουν στην αγορά. Η ε, λανθασμένη διαχείριση της γης σημαίνει ότι παράγουμε μόνο 40% αυτού που θα μπορούσαμε να παράγουμε. Αυτό είναι παράλογη κατάσταση. Αυτή η υψηλή, υψηλής έντασης μορφή εκμετάλλευση του πλανήτη μας δημιουργεί προβλήματα και στα υδάτινα περιβάλλοντα και δημιουργεί προβλήματα την υγεία των, υδα... Ε, υδάτων. Έχουμε για παράδειγμα τον ευτροφισμό των ε, φυκιών. Δημιουργούνται νεκρές ζώνες όπου δεν μπορούν να ζήσουν τα ψάρια. Γιατί δεν υπάρχει επαρκές ε, οξυγόνο. Μελέτες του 2004 αναφέρουν ότι υπάρχουν 140 τέτοιες νεκρές ζώνες στον κόσμο, οι μεγαλύτερη και πιο γνωστή είναι αυτή που συμβαίνει ετησίως στον κόλπο του Μεξικού λόγω των επιπτώσεων από τις ζώνες δημητριακών, καλλιέργειας δημητριακών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2002 αυτή η νεκρή ζώνη στον Ατλαντικό ε, ήταν περίπου όσο και η Μασαχουσέτη. Πρέπει να πω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αυτό που διαβάσαμε σε μια μελέτη στην Δανία όπου λέγεται ότι ο συνδυασμός από υψηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακος μπορεί να οδηγήσει αυτές οι νεκρές ζώνες που είναι τώρα γύρω στο 2% των υδάτων να είναι πάνω από 20% το 2100. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 25% του διοξίδιου του άνθρακα που εκλείουμε απορροφάται από τους ωκεανούς. Αλλά από ό,τι φαίνεται η δυνατότητα των ωκεανών να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο μειώνεται λόγω της ε, απώλειας των ε, οικοσυστημάτων στα παράλια. Για παράδειγμα, 13,5 γιγατόνι διοξίδιου του άνθρακα θα εκλειθούν ε, στην ατμόσφαιρα τα επόμενα 50 χρόνια λόγω του ότι η καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων στις παραλίες που υπήρξε μεταξύ του 1980 και του 2005 είναι τόσο μεγάλη και προκλήθηκε κυρίως από τις υδατοκαλλιέργειες. Αυτό είναι ισοδύναμο με όλες τις εκπομπές των 27, ετών, ε, των 27 χωρών συγγνώμη, της Ένωσης μεταξύ 1997 και 2005. Και επίσης έχουμε βέβαια υπεραλίευση, αλλαγή του κλίματος, τοξική μόλυνση, επιθετικά είδη και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και βιοτόπων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση συνολική και προληπτική για να διαχειριστούμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα ούτως ώστε να συνεχίσουμε να αντλούμε πλέον εκτήματα από την αλία καταλαβαίνοντας επίσης ότι η Γεωργία θα πρέπει να μας βοηθήσει να αναπληρώσουμε το έλλειμμα πρωτεϊνών που θα προκληθεί από τη μείωση των αλλιευμάτων. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνος όταν τονίζω ότι παρά το ότι δίνουμε 16 δισεκατομμύρια δολάρια δημόσιους πόρους κάθε χρόνο ως επιδοτήσεις, παρόλα αυτά κινδυνεύει η ε, θαλάσσια αλληλεία να, κατα... να καταγραμματιστεί. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό για πολύ καιρό. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα, αλλά ίσως αυτό να είναι και μια δυνατότητα επίλυσης που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες περιοχές. Η έρευνα στον τομέα αυτό, στον τομέα του ερυθρού τόνου του Βόρειου Ανατολικού Ατλαντικού, Εκτιμά ότι οι επιδοτήσει τη τάξη των 120 εκατομμυρίων δολαρίων αποδίδουν ένα ετήσιο κέρδο γύρω στα 70 εκατομμύρια δολάρια. Η έρευνα βρήκε επίση ότι η ε, αηφόρο μέλλον για την αλληλεία, ακόμα και χωρί επιδοτήσει, θα μπορούσε να παράγει ε, ετήσια κέρδη τη τάξη των 310 εκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος, εάν τα αποθέματα του τόνου θα μπορούσαν να επανέλθουν σε αηφόρο επίπεδο. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι εάν μπορούσαμε να εξαλείψουμε τα παρά, τις παράλογες επιδοτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να καταργήσουμε την υπερβολική αλληλεία, τότε θα μπορούσε η διεθνής αλληλευτική βιομηχανία να συμβάλλει με 250 δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος στον παγκόσμιο ΕΠ και αυτό σε αηφόρο βάση. Αυτό μας προσφέρει ελπίδες για μια θεραπεία μακροπρόθεσμη και όχι μια ανακούφιση πρόθεσμη και μια λύση που θα είναι προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων. Θα ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι ξέρω ότι η εφαρμογή των διαφόρων αποφάσεων και των δυσκό... είναι πολύ δύσκολη, αλλά αν σήμερα ξεχάσουμε να κοιτάμε το εδώ και τώρα και να κοιτάξουμε το μέλλον, δεν ξέρω αν έχουμε εναλλακτική λύση. Κυρίε και κύριοι, ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Κατά βάση, αυτό που, που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα σήμερα για να αποφύγουμε καταστροφές αύριο. Και μόνο τρόπο για να το κάνουμε αυτό είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, εστιάζουμε την προσέγγιση μας στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εάν τα αγροτικά και θαλάσσια συστήματά μας θα πρέπει να, να αντέξουν στον χρόνο, μακροπρόθεσμα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε σε κάθε τομέα πολιτικές που θα παρουσιάζουν σε πρώτη γραμμή το πραγματικό περιβαλλοντολογικό κόστος της καταστροφής περιβαλλοντολογικής και της καταστροφής του φυσικού κεφαλαίου. Έχω εξετάσει τα θέματα αυτά εδώ και 30 έτη και είχα την ευκαιρία να μπορέσω να έρθω σε επαφή με πάρα πολλούς καλούς καταπληκτικούς εμπειρογνώμονες και αναρωτιέμαι Εάν θα μπορούσα να σα παρουσιάσω μερικέ από μου, πώ πιστεύω θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε θα ήθελα να προτείνω ότι η κοινωνικονομική σταθερότητα βασίζεται στην αξία που δίδεται και στην υποστήριξη που δίνεται στις τοπικές κοινωνίες, στις παραδόσεις τους, αναγνωρίζοντας την συμβολή τους για την ανάπτυξη αναγνωρίζοντας τη συμβολή που παραδείγματος χάρη διαφορετικά συστήματα ε, αλίας προσφέρουν στην ε, δυνατότητα αυτή. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικά, διαφορετικά ε, αποτελέσματα όχι μόνο στην γεωργία αλλά και στον τουρισμό, στην ε, δασοκομεία και στη βιομηχανία. Και πιστεύω ότι χρειάζεται να έχουμε πολιτικές οι οποίες ενδυναμώνουν την κοινομορφία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ωφελήσουμε την ε, δημόσια οικονομία με το να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να προωθήσουμε ευφυείς επιδοτήσεις. Ο στόχος θα ήταν να ε, εστιαστούμε σε μια ποικιλομορφία της παραγωγής πιο συγκεκριμένα, προστατεύοντας όμως το δημόσιο καλό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν ενδυναμώσουμε την αντοχή της γεωργίας, ε, της γεωργίας ε, των θαλασσίων συστημάτων και των ενεργειακών συστημάτων για να είμαστε σίγουροι για την, για την ε, τροφοδότησή μας και θα αντέξουμε έτσι τα ε, ξαφνικά σοκ στις διεθνείς αγορές. Μπορούσαμε να έχουμε και μια διαφορετική προσέγγιση κέρδους και απολύων που θα μπορούσε έτσι να προωθήσει την κοινωνική και περιβαλλοντολογική ε, υπευθυνότητα των επιχειρήσεων και θα μας έδινε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις πράξεις μας καλύτερα. Και αυτό ακριβώς με έκανε να καθορίσω ένα σχέδιο της ε, της βιώσιμης ε, λογιστικής. Ε, ο στόχος ήταν να υπάρχει μια νέα προσέγγιση στην επιχείρηση, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ε, στοιχεία ε, στην, απόδοση μιας επιχειρήσης και χαίρομαι που ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων συμπεριλαμβαμένων της Βρετανικής κυβέρνησης και διεθνών ε, επιχειρήσεων όπως η DEDF, η HSBC, η Aviva υιοθετούν αυτό το σύστημα της ολοκληρωμένης λογιστικής. Πράγματι πέρσι διέβαινε το σχέδιο αυτό ξεκινώντας μια διεθνή ομάδα που θα στηρίζεται από, πολλούς, πολλά σώματα λογιστικής και καθορισμού προτύπων του κόσμου, καθώς επίσης και πολλές άλλες εταιρείες λογιστικής, διεθνής, τα χρηματοστήρια και το Ηνωμένα Έθνη. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι αυτή η πρωτοβουλία προέτρεξε των αποτελεσμάτων μιας μελέτης του Ηνωμένου Εθνών για την οικονομική οικοσυστημάτων και βιοποικιλομορφίας, TEEB, η οποία ε, παρουσίασε τα αποτέλεσματά της το περασμένο καλοκαίρι σε 193 υπουργούς περιβάλλοντος στην Αγκόγια. Έχοντας κάνει μία αξιολόγηση ε, της τάξης των πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομία όλου του κόσμου συμπεριλάμβανε και στοιχεία όπως την υγεία του φυσικού κεφαλαίου και αντικατοπτρίζει σωστά πώς οι υπηρεσίε που προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα αποδίδουν. Καθορίζοντας κάθε νέο πλαίσιο, οπωσδήποτε, υπάρχει και η ανάγκη να υπάρχει ολοκληρωμένη μορφή πολιτικών και μέσων μακροπρόθεσμης ε, πολιτικής για να ενθαρρυνθεί μια πράσινη οικονομία. Αυτή η οικονομία θα βασίζεται στη διαχείριση αηφόρων ε, μέσων καλύτερη ε, και πιο επικοδομητική επεξεργασία των απορριμμάτων, η κατασκευή νέων κτηρίων που δεν καταναλώνουν καθόλου ε, άνθρακα και η επίτευξη αυστηρής οικονομίας ενέργειας για τα κτίρια, τα αυτοκίνητα και τα αγαθά οικοκυριών. Εάν θα μπορούσαμε να εξετάσουμε όλο τον κόσμο κάτω από αυτή τη νέα οπτική γωνία, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια οικονομία η οποία αφενός θα τονίζει ακόμα περισσότερο στον προγραμματισμό αηφόρων αστικών εξέλιξεων και βοηθώντας τις ε, υπηρεσίες να διατηρήσουν την ποικιλομορφία και να εξασφαλίσουν τα οικοσυστήματα. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν θα βασίζονται τόσο πολύ σε κυβερνητικέ ε, επιδοτήσεις και εκείνους τους μηχανισμούς οι οποίοι περιέργως καταλήγουν στο να υποσκάπτουν το ζωτικό φυσικό παράγοντα που μας ε, ε, προσφέρουν τα ε, που μας προσφέρουν τα, τα οικοσυστήματα που έχουμε. Για να βρούμε τις λύσεις αυτές και να μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μια κλίμακα που θα είναι η πιο κατάλληλη, θα πρέπει να δούμε να υπάρχουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και θα χρειάζεται επίσης η γνώση πολλών εμπειρογνωμόνων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν θα μπορούμε να τα αφήσουμε όλα στην αγορά μόνο. Οι πολιτικές του δημοσίου τομέα θα πρέπει να είναι συνεπείς για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το απαραίτητο περιβάλλον στο οποίο θα μπορεί ο ιδιωτικό τομέα να επενδύσει. Μόνο τότε ο ιδιωτικό τομέα θα δεσμεύσει ε, κεφάλαια επιχειρηματικά. Η αγορά οπωσδήποτε προσφέρει μια δυνατότητα επιτάχυνσης αλλαγών στην συμπεριφορά. Αλλά για να είναι πραγματικά αποτελεσματικές, οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να εστιαστούν και να κατευθυνθούν ξεκάθαρα από μακροπρόθεσμες πολιτικές. Και αυτό σημαίνει αυστηρή νομοθεσία και, εάν μπορώ να το πω, επίσης αυστηρή εφαρμογή. Σε αυτόν τον κατάλογο θα ήθελα να προσθέσω μόνο μία πολύ σημαντική, ε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό είναι ο ρόλος του καταναλωτή. Νομίζω ότι εμεί ως καταναλωτές αρχίζουμε να ζητάμε αηφόρα προϊόντα και υπηρεσίες από τις υπηρεσίε και από τις κυβερνήσεις. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε οι νομοθέτες θα αρχίσουν να προσπαθούν να εισαγάγουν αυτές τις αλλαγές. Τελευταία αναρωτήθηκα γιατί ε, οι πολίτες δεν έχουν υιοθετήσει τις, τα πολλά πλεονεκτήματα για την προώθηση ενός ανηφόρου μέλλοντος. Το συμπέρασμά μου είναι ότι για πάρα πολύ καιρό οι περιβαλλοντολόγοι έτειναν να συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε αυτά που θα πρέπει οι πολίτες να σταματήσουν να κάνουν. Εάν συνεχώς λέγαμε ότι το να ζει κανένα ζωή φιλική προς το περιβάλλον σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει όλα αυτά που κάνουν τη ζωή αξιόλογη, τότε βέβαια όλοι θα αρνηθούν να αλλάξουν. Γι' αυτό ξεκίνησα μια νέα πρωτοβουλία που λέγεται STAR, αρχή δηλαδή, που έχει σαν στόχο να δείξει στους πολίτες αυτό που θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν. Μικρά βήματα για να μπορέσουμε να εκμεταλλευόμαστε καλύτερα τις φυσικούς πόρους μας. Συνεργαζόμενο με κάποιες από τις κύριες εταιρείες της Ευρώπης, Kingfisher, Eurostar, διακεκριμένα άτομα, ε, εμπειρογνώμες και επαγγελματίες του μάρκετινγκ, προσπαθούμε να πουλήσουμε, αν θέλετε, τα πλεονέκτηματα της αηφορίας. Όπως το είπε, μου είπε κάποιος, ε, εμπειρογνώμες του μάρκετινγκ, πρέπει να κάνουμε να είναι πραγματικά μοντέρνο, είναι cool, να χρησιμοποιεί κανείς λιγότερο υλικά, λιγότερα πράγματα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτή η προσέγγιση είναι πάρα πολύ θετική και προ όφελο των επιχειρήσεων, όπω ε, ανακάλυψε η Ματ Σπένσερ, μπορούν έτσι να κάνουν οικονομίε. Βέβαια, αυτή η διαδικασία δεν ε, βοηθήθηκε από την ε, πολύ αρνητική επίδραση της κοινή γνώμης εκείνων των σκεπτικιστών που θεωρούν ότι πρέπει πραγματικά δεν μπορεί κανένας να πιστεύει ότι οι κλιματολογικές αλλαγές οφείλονται σε ανθρώπινη βιομηχανική δραστηριότητα. Προτείνουν ότι εκατοντάδες εμπειρογνωμόνων γύρω από τον κόσμο και εκείνοι που δέχονται αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν ίσως να, είναι, να, μην έχουν μια αντικειμενική άποψη. Αναρωτιέμαι όμως γιατί ορισμένοι υποτίθεται ότι προσπαθούν να υποσκάψουν το σύστημα που βασίζεται στην αγορά, το καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα αντιμετωπίσουν τα εγγόνια τους και να τους πούνε ότι πραγματικά έχουν απετύχει όσον αφορά το μέλλον αυτών. Ότι αγνώρισαν όλες τις καθαρές και ξεκάθαρες προειδοποιήσεις λέγοντας ότι αυτό είναι μια κυκλική διαδικασία η οποία έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και που δεν μπορούσαν να ελέγξουν ότι αρνήθηκαν να ακούσουν τις απελπισμένες κραυγές εκείνων των τελευταίων παραδοσιακών κοινωνιών στον κόσμο που προειδοποιούσαν συνεπώς, συνεπώς για καταστροφές γιατί εκείνοι μπορούσαν να καταλάβουν τα μηνύματα της ε, επικείμενης καταστροφής στις έντονες διακυμάνσεις του συνήθως ε, αρμονικού ε, σχεδίου της φύσης. Αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν πραγματικά να αναλάβουν την ευθύνη που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση. Γιατί με αυτό το παιχνίδι παίζουν ρουλέτα με το μέλλον εκείνο που θα έρθει μετά από μας. Ένα μέλλον, μια κληρονομιά που θα καθοριστεί από αυτό που εσείς κυρίες και κύριοι θα αποφασίσετε εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, ε, δείξατε πολύ υπομονή να με ακούσετε. Σα ε, υπόσχομαι ότι αυτό που θα αποφασίσετε εδώ θα μπορέσει να οδηγήσει να ξεκινήσουν οι πολύ απαραίτητε προσαρμογέ που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θα ήθελα να σα ρωτήσω κατά πόσον θα έχετε την τόλμη να δράξετε τη ευκαιρία, να ορίσετε, να καθορίσετε για την Ευρώπη μία οδό επιβίωσης και οικονομικής ευμάρειας και έτσι να κερδίσετε την ευγνωμοσύνη των απογόνων μας. Uh, Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι δώσατε ορισμού σε πολλά από τα σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Συνδέσατε το κλίμα με την ενέργεια, με τα τρόφιμα, με το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι δύσκολα προβλήματα και είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα, δεν έχουμε προπαρασκευαστεί πλήρως για να χρηματοδοτήσουμε όλες τις προσπάθειες και να κάνουμε τα βήματα προς την αποτελεσματικότητα και προς την εξοικονόμηση ενέργειας που είναι απαραίτητα και στα πλαίσια της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί αν δεν υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε και πολλά στον συγκεκριμένο τομέα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ σημαντική σας ομιλία. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Σοζέ Μανουέλ Μπαρόσο. Your Royal Ψηλότητά σας, κύριοι κύριοι πρόεδροι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι προσκεκλημένοι. Πραγματικά αυτή η συνάντηση είναι έκτακτη. Σπάνια να βλέπει κανείς τέτοιες συναντήσεις υψηλού επίπεδου ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εξοχότητά σας για μια πάρα πολύ πυκνή και σημαντική για όλους μας ομιλία. Αυτή η εταιρική σχέση νομίζω είναι απαραίτητη για να οδηγηθούμε στην αηφορία. Είμαι ευγνώμων λοιπόν στο πρόγραμμα Cambridge του Πρόεδρου Μπούζεκ και της αυτοεξοχότητος έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αυτήν εδώ τη συνάντηση σήμερα. Και ο τίτλος αυτής εδώ της συνάντησης «Ευημερία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών» κάτι δείχνει. Η συνέργεια ανάμεσα στις χαμηλές εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και την πρόοδο θα μας οδηγήσουν στην πραγματική αηφορία στην ανάπτυξη που όλοι επιθυμούμε. Όταν μιλάμε για την οικονομία με χαμηλές εκπομπές και την αποτελεσματικότητα της ενέργειας δεν τα κάνουμε αυτά για να φανούμε της μόδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι αυτά θα μας οδηγήσουν σε μια πραγματική ανάπτυξη η οποία δεν είναι μέσω αυτών των προσπαθειών κάποια επιλογή αλλά είναι απαραίτητο έτσι ώστε να τοποθετήσουμε την Ευρώπη σε σωστή πλεονεκτική θέση για το 2020 δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. Εδώ και λίγες εβδομάδες πήραμε τη λεγόμενη βασική πρωτοβουλία θα έλεγα για την Ευρώπη του 2020 έτσι μόνο θα μπορέσουμε να διασώσουμε τον πλανήτη, να διασφαλίσουμε τις προμήθειες τις οποίες έχουμε ανάγκη και να αναπτυχθούμε οικονομικά χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τους πόρους. Τρεις προϋποθέσεις νομίζω είναι απαραίτητες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρώτον, απαιτούνται επιμέρους δράσεις σε πάρα πολλούς τομείς με συγκεκριμένο πολιτικό βάρος και υποστήριξη από το κοινό και από τον επιχειρηματικό κόσμο έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν όλοι την προσπάθεια αυτή. Η αποτελεσματικότητα των πόρων δεν μπορεί να περιοριστεί στο λεγόμενο πρασίνισμα σε εισαγωγικά των διαδικασιών, αλλά μια καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις θα τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές σταθερές, αναπτυξιακές και μακροπρόθεσμες. Θα ενθαρρύνει επίσης και τους καταναλωτές να κάνουν αντικαταστάσεις στους τρόπους με τους οποίους καταναλώνουν έτσι ώστε να μην εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι. Οι προσπάθειες μας αυτές για την αποτελεσματικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων είναι ο κοινό παρανομαστής και στον τομέα της γεωργίας και στον τομέα της αλίας και στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της διαχείρισης της ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα είναι ξεκάθαρα. Καλύτερη οικονομική απόδοση, μείωση των φυσικών πόρων, εντοπισμός νέων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την καινοτομία, διασφάλιση των προμηθειών των φυσικών πόρων τη στιγμή κατά την οποία ο ανταγωνισμός για την κατανάλωση των πόρων αυτών αυξάνεται, κατά πολέμηση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών και πολέμηση φυσικά της σπατάλης στους φυσικούς πόρους. Αυτό θα πρέπει να περάσει σαν λογική και στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, σε καλύτερη κατανόηση του τρόπου που καταναλώνουμε. Κάποιες δράσεις απαιτούν όμως σημαντικές επενδύσεις και τεχνολογικές βελτιώσεις και σημαντικές ε, μεταβατικές περιόδους, ιδιαίτερα σε συστήματα μεταφορών και κατανάλωσης. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν εν μία νυχτή. Αλλά δεν θα συμβούν ποτέ αν οι επιχειρήσεις δεν είναι απόλυτα σίγουρες για να μπορέσουν να επενδύσουν έτσι ώστε οι μελλοντικέ γενιές να ωφεληθούν από αυτές τις έξυπνες επενδύσεις. Ένα διακανονιστικό πλαίσιο θα παράσχει νομίζω αυτή τη βεβαιότητα. Πρέπει να βοηθήσουμε να επενδύσουμε στους επιστήμονές μας την έρευνα και τότε και οι επιχειρήσεις θα μας βοηθήσουν να αναζωογονήσουμε τα κέντρα των πόλεων, να καταπολεμήσουμε την τοξική βροχή και υπάρχουν ενθαρρυντικά θα έλεγα σημεία για όσους ε, πράγματι επιθυμούν να δουν την αλήθεια. Από το 1990 μειώσαμε τις εκπομπές καυσαερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 10% ενώ οι οικονομίες μας αυξήθηκαν κατά 40%. Μειώνουμε επίσης την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και δημιουργούμε εναλλακτικέ λύσεις. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σαν παράδειγμα. Από τα 25 μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, τα 23 από τα 25 βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να επεκταθούν και σε άλλους τομείς έτσι ώστε να εφελθούν όλοι. Η επιτυχή στρατηγική οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής γενικότερα. Θέσεις εργασίας στον τομέα της αηφορίας σαν παράδειγμα είναι σταθερές θέσεις εργασίας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Οι νέες τεχνολογίες ε, βοηθούν στη μείωση των εκπομπών καυστέριων και βελτιώνουν τη δημόσια υγεία. Αυστηρότεροι κανόνες στον τομέα του περιβάλλοντος οδηγούν σε νέα κίνητρα στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και έρευνες έχουν δείξει ότι διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφορούν κυρίως πλέον ε, την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων ιδιαίτερα μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας του Κιώτο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ψευδεστήσεις, οι άλλες περιοχές του κόσμου πηγαίνουν γρήγορα και κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πλεονεκτήματα τα οποία είχαμε σε κομβικούς τομείς. Στην Άνοιξη θα πάρουμε τις τελικές αποφάσεις έτσι ώστε να μειώσουμε ε, τις εκπομπές καυσαερίων μέχρι το 2050 κατά 80 με 90%. Ταυτόχρονα θα παρουσιάσουμε και το όραμα το οποίο έχουμε για, μια, για ένα ανταγωνιστικό και αηφόρο και οικονομικό σε κατανάλωση ενέργεια σύστημα μεταφορών μέχρι το 2015. Έτσι θα μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας κατά 20% και νομίζω θα τα συνδυάσουμε αυτά και με τα επιτυχημένα αποτελέσματα του Συμβουλίου Κορυφής της προηγούμενης Παρασκευής. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποσυνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη από την χρήση των φυσικών πόρων Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και τις πρώτες μελέτες προς την κατεύθυνση αυτή ήδη μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και θα επηρεάσουν και την κοινή αγροτική πολιτική και την αλλιευτική πολιτική και όλα αυτά θα διαμορφώσουν τις συνθήκες έτσι ώστε και μέσω του προϋπολογισμού του 2012 να βελτιωθούν τα πράγματα και θα τεθεί το θέμα επίσης και της φορολόγησης στον τομέα αυτό. 2,5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, θα οδηγείται μάλλον και καλύπτει ακριβώς την προμήθεια ενέργειας και πολλές από τις θέσεις απασχόλησης άνω των 2 εκατομμυρίων εξαρτώνται από το συγκεκριμένο τομέα. Αυτό το οποίο λοιπόν συζητάμε εδώ είναι στην ουσία ένας αγώνας εναντίον του χρόνου. Τα βήματα τα οποία προτείνουμε δεν είναι βήματα προς τα πίσω όπως λένε ορισμένοι. Αντίθετα δημιουργούμε ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι φιλικό για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Οι προσπάθειές μας θα οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Θεωρώ ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς οι οποίοι καταλωνούν ότι το να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα είναι δύσκολο μεν αλλά και είναι και το πιο επιτυχές. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολλά μέσα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι η πολιτική βούληση και οι εταιρικέ σχέσεις. Και αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι επιθυμία για συνεργασία υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μπαρόζο, για την ομιλία σας και για την απολυσματικότητα σας στην ε, προετοιμασία σα και στην περασμένη θητεία και στην τρέχουσα. Προετοιμάστε, λέω, όλα τα σχέδια νομοθεσία που έχουν σαν στόχο όχι μόνο την κοινή ενεργειακή πολιτική, αλλά καταρχήν την ε, προστασία του κλίματος ε, για να κινηθούμε προς ένα περιβάλλον φιλικό προς εξελίξει. Επόμενο ομιλητή, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Σέμαν Φων Ρόμπεϊ. Ευχαριστώ. Υψηλότατε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιότιμα μέλη, ε, κυρίε και κύριοι. Η απόφαση σα να εστιάσετε τη σημερινή συζήτηση στην οικονομία χαμηλή κατανάλωση άνθρακα είναι πάρα πολύ επίκαιρη μέσα στα πλαίσια Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 27 αρχικών κρατών και κυβερνήσεων, αφιέρωσε ένα μεγάλο τμήμα της συνεδρίασής του στο θέμα της ενέργειας. Πρώτη φορά που εργοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν το θέμα αυτό σε τόσες λεπτομέρειες. Καταδεικνύει αυτό μια προσωπική δέσμευση στο επίπεδο αυτό που είναι ουσιαστική για να υπάρξουν αποτέλεσμα και στο επίπεδο Ένωσης και στο επίπεδο κρατών μελών. Όσον αφορά την ανάγκη ενέργειας χαμηλής κατανόλωσης ε, άνθρακα ελεγχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα προωθήσουν επενδύσεις για αηφόρα ενέργεια με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Ο στόχος του να μειωθούν οι εκπομπές ε, του, ε, του θερμοκηπίου μέχρι το 1950 κατά 80-85% θα απαιτήσει επανάσταση στα ενεργειακά συστήματα. Επανάσταση που πρέπει να αρχίσει σήμερα. Σημαίνει αυτό μία νέα βιομηχανική επανάσταση. Οι αποφάσεις της σήμερα θα καθορίσουν τα σύμβολα της αύριο. Όλα αυτά θα απαιτήσουν επενδύσεις. Επενδύσεις σε λύσεις για ε, εξοικονόμηση ενέργειας για τις πόλεις, ανάπτυξη καηφόρων βιοκαυσίμων και στην ανάπτυξη καθαρών οχημάτων. Εφαρμογή της οδηγίας για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα υποστήριξης, θα είναι ουσιαστικά. Κυρίως, οι επενδύσεις στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι πάρα πολύ ουσιαστικές αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, υποστηρίζουν την ασφάλεια στην τροφοδότηση, μειώνουν ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι απλό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια. Ας μην ξεχάσουμε μια απλή λογική ότι η πιο φτηνή και η πιο πράσινη ενέργεια είναι εκείνη που δεν χρησιμοποιούμε. Η στόχη αποτελεσματικότητα για το 2020 που αποφασίστηκε τον Ιούνιο στο, Συμβούλιο ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ακολουθεί την σωστή οδό αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να επιτεχυνθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι δυνατότητε εξοικονόμηση ενέργεια που υπάρχουν στα κτίρια, στι μεταφορέ και στι διαδικασίε. Ε, από την 1η Ιουνιού του επόμενου έτου, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα πρότυπα ε, αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας στις δημόσιες αγορές και στα δημόσια κτίρια. Και θα υπάρξει και μια πρόταση Κομισιόν για ένα νέο σχέδιο για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα που θα καθορίζει νέους στόχους, πολιτικές και μέτρα για όλη την αλυσίδα της τροφοδότης ενέργειας. Περισσότερες τεχνολογίες που θα, που θα χρησιμοποιούμε γι' αυτό δεν υπάρχουν ακόμα. Χρειάζονται λοιπόν υποστήριξη για την ανάπτυξή τους και την εφαρμογή τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο καλεί να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα μικρά δίκτυα μέχρι το 2012. Και αυτό επίσης τα θέματα της ένταξης στο δίκτυο των ε, ε, μονάδων παραγωγής αιωλικής ενέργειας. Σημαίνει αυτό ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε την δημόσια αποδοχή ορισμένων θεμάτων. Παραδείγματος χάρη ορισμένες μορφές ε, ανανεώσιμης ενέργειας και επίσης η υπόγεια αποθήκευση του διοξείδου του άνθρακα. Πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα. Αυτό χρειάζεται κατεπηγόντως και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους. Θα πρέπει να έχουμε ασφαλή, αηφόρα και φτηνή ενέργεια που θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αυτό παραμένει ένα κύριο θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει προστιθέμενη αξία σε αυτούς τους στόχους. Στο παρελθόν πολλές προσπάθειες κατεβλήθησαν για τις κύριες πολιτικές ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη οδηγίες για την ενέργεια, για τις κλιματικές αλλαγές και οποιαδήποτε δευτερεύουσα νομοθεσία υποστηρίζει τους στόχους αυτούς. Τη περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την δέσμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους στόχους αυτούς και κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα πετύχαμε την προσωπική πολιτική δέσμευση των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν προτεραιότητα στους στόχους αυτούς. Αυτό σημαίνει να συνδυάσουν αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένα ξεχωριστά στη χώρα μα με αυτό που μπορούμε να κάνουμε από κοινό. Να πετύχουμε έτσι συνέργειε και, οικονομικές, ε, και οικονομίε κλίμακα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πρώτα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η μεγαλύτερη νέα αγορά του κόσμου, θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη δική μας Ήπειρο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μας στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα προσεκτικής αισιοδοξία παρόλο που δεν είναι πολιτικά σωστό να είναι κανένα αισιόδοξο. Στην Ευρώπη εμεί μπορούμε να καθορίσουμε φιλόδοξους στόχους πολλές φορές πριν από το υπόλοιπο κόσμο και να ε, ε αναλάβουμε ευθύνες για να οδηγηθούμε και σε αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε όμως την ενίσχυσή σα Γι' αυτό μια διάσκεψη όπω αυτή σήμερα, η δική σα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί βλέπω ότι ενώνονται εδώ ορισμένοι από τους διεθνείς εμπειρογνώμονες ε, που ε, είναι ηγέτες στον τομέα αυτό, καθώς επίσης και τους νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προβλέπω να ακούσω τις ιδέες που θα απορρέουν από τη σημερινή συναντήση και να δούμε τι μπορεί να γίνει από εσά. Εξετάζοντας το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον, που είναι η μου, δική μου φιλοδεξία ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορείτε να περιμένετε λιγότερο από ένα μόνιμο πρόεδρο, Έχω να πω ότι δεν υπάρχουν πολλά πιο σημαντικά θέματα από εκείνο που εξετάζετε εσείς σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την εργασία σας και να ευχαριστήσω την υψηλότητά σας ε, για την παρουσία σας εδώ που δίνει ιδιαίτερη ε, σημασία στη δική μας προσπάθεια. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Mr. President, for... Ευχαριστώ, Πρόεδρε για την παρουσίασή σας και τις παρατηρήσεις σας και για την οργάνωση της τελευταίας συνάντησης του Συμβουλίου. Δεν πετύχαμε όσα θα θέλαμε βέβαια. Αλλά και αυτό το, αυτή η συνάντηση ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί αποδεικνύει το ενδιαφέρον που έχουμε γενικότερα για τα θέματα αυτά. Γι' αυτού εξοχότης πρέπει να φύγει λοιπόν πλέον, να αποχωρήσει η εμπλοκή σας στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εξοχότητά σας και για την παρουσίασή σας και τις ιδέες τις οποίες θέσαμε, οι οποίες είναι καθοριστικές για μας. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία συζητούμε συστηματικά και μέχρι τώρα δεν έχουμε πετύχει ό,τι θα επιθυμούσαμε να πετύχουμε εδώ και 5 με 7 χρόνια. Αλλά σημειώθηκε πρόοδος. Σημαντική πρόοδος. Απαιτούμε την εμπλοκή μας και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για θέματα κλίματος και η παρουσία σας εδώ, η υποστήριξή σας και αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να ζούμε σε ένα περιβάλλον φιλικό για τη φύση και τον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. It uh, intervention, the Τώρα θα ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση με την κυρία Κορίν Λεπάζ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφαλείας Τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε τρία λεπτά, χρόνο ρεκόρ, θα πρέπει να κάνω την εισαγωγή της ε, όλης συζήτησης μετά από τις τόσο σημαντικές τοποθετήσεις που ακούσαμε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτο, το να έχουμε φιλόδοξους στόχους στο ύψος των προκλήσεων. Όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι, όποιος και, όποια και να είναι η θέση μας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Πρέπει να είμαστε περήφανοι διότι είμαστε η μόνη περιοχή στον κόσμο η οποία έθεσε τόσο υψηλούς στόχους. Αλλά και η εξοχότης του μας το θύμισε, οι στόχοι είναι πάρα πολύ ψηλοί. Και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη σημαντικές. Εγώ με τον ενθουσιασμό των χωρών του Νότου λέω ότι άμα, πρέπει να, θέλουμε να κρατήσουμε τον κυριαρχικό μας ρόλο στον τεχνολογικό τομέα θα πρέ... και τον βιομηχανικό τομέα θα πρέπει να θέσουμε υψηλότερους στόχους και για τις εκπομπές του θερμοκηπίου αλλά και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα από την άλλη. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να ντοπάρουμε την βιομηχανία μας για να μπορέσει να κρατήσει τον ηγετικό της ρόλο. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι το να έχουμε συνεκτικούς στόχους μέσα στις πολιτικές καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και συνεκτικούς στόχους και μεταξύ των διαφόρων πολιτικών μας στο εσωτερικό της καταπολέμησης, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος είναι απαραίτητο αν πρέπει να έχουμε ένα σύστημα ποσοστώσεων που λειτουργούν εύρυθμα αν θέλουμε μια πραγματική αποδοτικότητα των επενδύσεών μας που θα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε στην ανάπτυξη ορυκτής, ε, βιομηχανίας ορυκτών. Δηλαδή στη βιομηχανία του σχιστόλιθου και άμμος που χρησιμοποιείται στην, για την ε, κατασκευή ασφάλτου. Δεν αξίζει τον κόπο εμείς να προσθέτουμε παραπάνω στην μόλυνση από το πετρέλαιο και αυτού του είδους τις επενδύσεις. Βέβαια άλλο είναι να το θέλουμε και άλλο είναι να σταματήσουν να σταματήσει η ενθάρρυνση αυτών των επενδύσεων. Τώρα εμείς μιλάμε για low carbon economy σήμερα. Αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Μήπως θα έπρεπε να μιλάμε για μία φτωχή σε απόβλητα οικονομία διότι οι εκπομπές άνθρακος και αυτές απόβλητα είναι αυτό θα μας επέτρεπε να έχουμε μια ολική αντίληψη και να κάνουμε και τις σωστές επιλογές και για, κυρίως ε, για τις ενέργειες, φτωχές εκπομπές ε, άνθρακος πρέπει να είναι αηφόρες και να μην οδηγούν στη δημιουργία αποβλήτων. Δεν μπορούμε εμείς να εξισώνουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πηγές ενέργειας φτωχές σε παραγωγή άνθρακα αλλά οι οποίες δημιουργούν απόβλητα. Και ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο κρατώντας τα τρία μου λεπτά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τα βάλουμε, να τα εντάξουμε όλα αυτά μέσα σε ένα νέο γενικότερο όραμα μέτρησης να αρχίσουμε να μετράμε διαφορετικά και να διαμορφώνουμε τις νέες μας πριωτερότητες, να βλέπουμε τις κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιλογών μας. Και έτσι θα μπορέσουμε εμείς να πετύχουμε την οικονομική ευημερία και να τη συνδέσουμε με το γενικότερο αίσθημα ευθυνών που έχουμε εμείς έναντι των μελλοντικών γενεών. Αυτά τα σύντομα εισαγωγικά. Κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θα ήθελα παρακαλώ να υπάρχουν σύντομε παρεμβάσει. Κύριε Χέρτσο, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ που οργάνωσατε τη διάσκεψη αυτή που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να καταστήσουμε κάθε τι δυνατό με τα, τις δυνατότητες που έχουμε για να προωθήσουμε την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συγγήτρια της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, και για τον προπολογισμό θα ήθελα να αρχίσω με κάτι που έμαθα από τη μητέρα μου όταν είμαι μικρή που έλεγε ότι το να έχει κανένα μια ιδέα δεν είναι η λύση, η λύση είναι η εκτέλεση. Η ιδέα μου λοιπόν είναι όταν έχουμε τον ενθουσιασμό των Ευρωπαίων πολιτών, αν έχουμε το όραμα των δικών μας ηγετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχουμε την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε μια τελευταία δέσμευση από τα κράτη-μέλη, δηλαδή αυτό δεν εντάχθηκε ούτε στο παλιό προπολογισμό ούτε στον τρέχοντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές για μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Η ερώτησή μου στρέφεται προς τον κύριο Βαν Ρομπόη. Μετά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ακούσαμε ότι τα προγράμματα, το στρατηγικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα το τεχνολογικό θεωρούνται σαν πολύ σημαντικά βήματα και σε σχέση με τις τεχνολογίες που χρειαζόμεθα και επίσης ε, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε καινοτομικές λύσεις. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα είναι πότε θα διαθέσουν τα χρήματα τα οποία έχουν υποσχεθεί τα κράτη-μέλη. Εδώ μπορείτε να μας απαντήσετε. Ο πρόεδρος Μπαρόσο. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη αλλά και εγώ έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση σε 8 λεπτά. Προσπαθώ να σεβαστώ το χρονοδιάγραμμα και δεν μπορώ να ακούσω το σύνολο της συζήτησης αλλά φυσικά η Επιτροπή παρακολουθεί τις συζητήσει σα και είναι ιδιαίτερο ευτυχή να επανέλθει στο Κοινοβούλιο και να συζητήσει τα θέματα αυτά εκ νέου μαζί σας. Να αντιδράσω λίγο στα σχόλια τα οποία ακούστηκαν. Πρώτον, να πω ότι όλοι ακούσαμε την αυτού εξοχότητα τον πρίγκιπα της Ουαλίας, ο οποίος ε, μας ενέπνευσε με την ομιλία του, αλλά και σε επίπεδο ουσίας μας ενέπνευσε. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το, αυτή την όθηση την οποία έχουμε ήδη δώσει στις συζητήσεις αυτές. Η υποστήριξη βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης ε, είναι θα έλεγα σε σχέση με αυτά τα προγράμματα πιο περιορισμένη από ό,τι πριν 2-3 χρόνια και η κυρία Χέρτσοκ και η κυρία Χέκ ουσιαστικά αναφέρθηκαν σε αυτά. Απαιτείται και δημόσια παρέμβαση και δημόσια επέμβαση ενώ εδώ ε, σε οικονομικό επίπεδο και γι' αυτό η συζήτηση χρειάζεται περαιτέρω όθηση και περαιτέρω συνειδητοποίηση της οξύτητας των προβλημάτων και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε όλα αυτά όχι μόνο την παρουσία ή την απουσία του ε, πρίγκιπος της Ουαλίας αλλά και φυσικά την παρουσία όλων των σημαντικών εμπειρογνωμόνων που είναι ανάμεσά μας σήμερα. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτά τα οποία συζητάμε δεν είναι σημαντικά μόνο σε επίπεδο περιβαλλοντικό και κλιματολογικό, κάτι το οποίο είναι έτσι και αλλιώς σημαντικό δραματικά, αλλά είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Είναι η κομβική θα έλεγα πολιτική απάντηση και για τα προβλήματα και τις απορίες τις οποίες έχουμε σχετικά με τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Θυμίζω ότι η διαδικασία αυτή είναι μια σφαιρική διαδικασία, δεν είναι κάτι το ευρωπαϊκό. Συζητάμε με τους φίλους μας, τους Αμερικανούς, αλλά και τις αναδυόμενες οικονομίες. Απαιτείται λοιπόν η συζήτηση αυτή να γίνει αντικείμενο διαχείρισης με τέτοιο τρόπο, με σωστό τρόπο, έτσι ώστε κανείς να μην αποκλειστεί, κανείς να μην εξαιρείται και να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να ζητάμε και από άλλους να σέβονται τις υποχρεώσεις μας αυτές και να αναλαμβάνουν αντίστοιχες. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι η συνάντηση, το Συμβούλιο το τελευταίο, νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση αυτή στον τομέα της αποτελεσματικότητας και της ενέργειας. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας. Θα μπορέσουμε, ελπίζω, να οδηγηθούμε στη μείωση κατά 20% των εκπομπών καυσαερίων μέχρι το 2020. Έχουμε κάνει κάποια βήματα θετικά, αλλά δεν είμαστε όμως σε σωστό δρόμο θα έλεγα για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και γι' αυτό εκεί πολλά μένει να γίνουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο προέδρους μας για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Περνάμε τώρα στις οικονομίες της ανταγωνιστικότητας και χαμηλής εκπομπής καυσαερίων. Είναι ο δεύτερος γύρος των συζητήσεων. Θα συνεχίσει να προεδρεύει ο συνάδελφος Ρολ, πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε δύο λεπτά θα ξεκινήσει η συζήτηση αυτή, ο νέος γύρος των συζητήσεων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 Sehr geehrte, Damen und Herren, και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, έχουμε ακόμα 40 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας. στο πάνελ αυτό να εμβαθύνουμε με υψηλή, υψηλού επίπεδου προγραμμάτων και θα πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι γιατί ε, θα πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο μας και θα πρέπει και οι συνάδελφοι να συνεχίσουν κατόπιν με τα άλλα θέματα συζήτηση. Ακούσαμε πάρα πολλά ουσιαστικά θέματα και έχουμε τώρα την ευκαιρία να έχουμε ε, τους επιρρογνώμενους εδώ με τη βοήθεια των οποίων θα εμβαθύνουμε κάποια από τα θέματα. Έχουμε μεταξύ μας τον Λόρδο Νικολά καθηγητή οικονομία και Διακυβέρνησης ε, στο Research Institute of Climate Change and the Environment στο London School of Economics. Ε, σας καλωσορίζω εδώ. Καλωσορίζω επίσης τον κύριο Γκάρατ Φόρ που είναι ο ε, Γενικός Διευθυντής του Philips Lightning MA και τον κύριο ο οποίος αντικαταστά τον κύριο Σουίνι από την Shell ο οποίος δυστυχώς αναγκάστηκε να ξαναφύγει γιατί σήμερα τη νύχτα είχε μια πολύ δυσάρεστη σύγκρουση σε έναν συνδρομικό σταθμό των Βρυξελών με εγκληματικά στοιχεία και αναγκάστηκε να φύγει κατεπηγόντως. Πρώτος έχει ο Λόρδος Νικολάς Σας παρακαλώ να μας αποτείνετε σύντομα το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας σε ε, μια τόσο σημαντική ευκαιρία. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά επίγουσες δράσεις θα πρέπει να γίνουν, αλλά και οι δράσεις αυτές είναι πολύ ελκυστικές. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι δεν είμαστε ακόμα αρκετά πιστικοί στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε και θα πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοσή μας συγκεντρώνοντας τα επιχειρήματα. Θα πρέπει καταρχήν να κατανοήσουμε ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικότατοι. Είναι υπαρξιακοί θα έλεγα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και του πλανήτη. Αν συνεχίσουμε όπως πάμε και συγκεντρώνονται έτσι τα, το διοξείδιο του άνθρακα και τα αέρια του ε, θερμοκηπίου, θα αυξηθούν μέχρι τα τέλη του αιώνα από 4,35 ppm σε 7,5 ppm. Δηλαδή θα έχουμε 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από αυτό που είχαμε τον, ε, τα μέσα του 19ου αιώνα. Εμείς είμαστε εδώ 200.000 έτη μόνο στον πλανήτη αυτό ως Homo sapiens και αυτή η στάση μας θα μετέτρεπε το που ζούμε και θα οδηγούσε στον θάνατο εκατομμυρίων, όχι δισεκατομμυρίων ανθρώπων και θα οδηγούσε σε συγκρούσεις παγκόσμιες. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Ως ανθρώπινα όντα δεν είδαμε πουθενά μια τέτοια ανάπτυξη της θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι λοιπόν το διακύβευμα. Τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ τα επιχείρηματα είναι πιο ελκυστικά. Κατά βάση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την κλίμακα των παράξεων που χρειάζονται, ώστε να έχουμε μια ευκαιρία έστω και 50% να μείνουμε σε μια αύξηση του δύο βαθμών. Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε κατά 50 δισεκατομμύρια από 50 δισεκατομμύρια τόνους εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα το έτος στις 20 περίπου, δηλαδή μία μείωση με να συντελεστεί 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή κατά 3 επί 2,5. 8 δηλαδή επειδή αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε παντού, αυτό σημαίνει ότι εκεί που μπορούμε να δράσουμε θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές στο μηδέν. Αυτό είναι μια ενεργειακή και βιομηχανική επανάσταση. Είναι μια επίπτωση της αριθμητικής που χρειάζεται. Τι είναι βέβαια προς μια βιομηχανική επανάσταση. Αλλά κοίταξε κανένα στις περασμένες βιομηχανικές ε, επαναστάσεις από την μηχανοποίηση τα τέλη του 18ου αιώνα και την τρέχουσα της ε, τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, αυτές οι βιομηχανικές ε, επαναστάσεις οδηγούν σε τρεις-τέσσερις ε, ε, δεκαετίες ανάπτυξης με τις επενδύσεις να αυξάνονται. Και θα πρέπει να ακούσουμε το πολύ σημαντικό μήνυμα στην Ευρώπη του τι πρέπει να κάνουμε. Και αν σκεφτούμε τι σημαίνει ανάπτυξη με χαμηλή κατανάλωση ε, άνθρακα, αυτό σημαίνει ότι είναι πιο ασφάλεια όσον αφορά τον άνθρακα, καθαρή, πιο ε, χαμηλότερους ε, θορύβους και οικονομική. Λοιπόν, ο στόχος είναι πολύ πιο ελκυστικός από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριβόμασταν σήμερα ή και στο παρελθόν. Βέβαια, ε, βιομηχανική επανάσταση σημαίνει μετατόπιση και σημαντικές επενδύσεις δεν είναι δωρεάν, αλλά είναι πολλά υποσχόμενη και ελκυστική δραστηριότητα. Πώς θα φτάσουμε εκεί, ποια είναι η μορφή της δράσης. Θα πω δύο λόγια για την δημόσια πολιτική και μετά τις δράσεις. Πολιτική σημαίνει ότι θα διορθώνονται οι αποτυχίες της αγοράς. Δηλαδή έτσι μπορεί η αγορά να λειτουργήσει σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε το εξωτερικό κόστος των ε, αερίων του θερμοκηπίου, γιατί αν δεν τους βάλουμε μία τιμή, δεν θα το αντιμετωπίσει κανένας. Ας το φτιάξουμε αυτό. Ανάπτυξη και έρευνα οδηγεί σε ωφέλη για άλλους και βιαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τα ωφέλη αυτά. Χρειαζόμαστε επίσης άλλοι να υιοθετήσουν αυτό που κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την έρευνα και εν ανάπτυξη. Επίσης, οι κεφαλαιογορές ξέρουμε ότι δεν αργώνται πάρα πολύ καλά όσον αφορά μακροπρόθεσμες επενδύσεις με υψηλό κίνδυνο. Και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Οι μεταφορές. Και εκεί υπάρχει ένα εξωτερικό κόστος πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μεγάλο δυναμικό της Νοτιού Ευρώπης για την ε, ηλιακή ενέργεια εάν δεν έχουμε καλύτερα ε, συστήματα δικτύων. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ε, προωθήσει η πολιτική. Παραδείγματος χάρη είναι ε, οι αγορές παραδείγματος χάρη πληροφόρησης θα πρέπει όλοι να είναι πολύ πιο καλά ενημέροι για το τι μπορούν να κάνουν. Πολύ μπορούν να βοηθήσουμε εδώ βέβαια ε, και όσον αφορά τις ε, ετικέτες που δίνονται στα προϊόντα κλπ. Αυτές είναι ορισμένες πολιτικές που χρειαζόμαστε για να δώσουμε ενάσματα στην οικονομία, στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σωστά και θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο αυστηρά στην Ευρώπη ώστε αυτές οι πολιτικές να είναι σαφείς, ισχυρές και προβλέψιμες. Κάνοντας αυτό, ξεκινάμε επενδύσεις οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει, αλλά θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ισχυρέ αν έχουν σαφείς και ισχυρε. Δημόσιε πολιτικές. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο υψηλή η τιμή του άνθρακα, πιο έντονη υποστήριξη από την Ευρώπη της έρευνας και της ανάπτυξης, που έχει μειωθεί κατά 50% από τη δεκαετία του 80 του περασμένου αιώνα. Δίχτυα, υποδομή και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και ε, εκπομπές από τις μεταφορές, όλα αυτά θα πρέπει να διακανοστούν. Πού θα πρέπει να δράσουμε. Νομοθετικά μέτρα είπα, αλλά σε ποιους τομείς. Σε όλους. Γεωργία, κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές, η ηλεκτρική ενέργεια. Εγώ πάντα θέτω την ηλεκτρική ενέργεια στο τέλος, γιατί οι περισσότεροι τη βάζουν μπροστά. Αλλά θα πρέπει να είναι παντού, παντού. Αυτή η βιομηχανική επανάσταση είναι επανάσταση για όλη την οικονομία και πολλά μπορούμε να κάνουμε. Καλύτερη γεωργία, καλύτερη, ε, ε, καλύτερη μόνωση των κτηρίων, ε, ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια κλπ. Πολλά πρέπει να γίνουν και παντού πρέπει να γίνουν, όχι ένα μόνο. Η βιομηχανική επανάσταση αυτή απασχολεί και την κοινότητα εκάστοτε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν βασιστεί στις κοινότητες. Όσο πιο πολύ εμπλακούν οι κοινότητες, τόσο πιο καλά θα α, εκτιμηθούν οι δράσεις. Συνεχώς υπάρχουν νέες ιδέες. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήμασταν πάρα πολύ δημιουργικοί. Τα κεφαλαια τώρα ρέουν σιγά σιγά, αλλά χρειάζεται περισσότερη δημόσια πολιτική, ούτως ώστε να φτάσουμε στην απαραίτητη κλίμακα που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι τροποποίησεις κλίμακας που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη με μικρή κατανάλωση άνθρακα είναι η πραγματική ανάπτυξη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, έχουμε μια καλή πολιτική. Η ανάπτυξη με υψηλή κατανάλωση ε, άνθρακα είναι μια αντίφαση γιατί θα αυτοκαταστραφεί. Ακαδημίκη σαν εμένα θα πρέπει να πούμε στους ε, βουλευτές ε, θα πρέπει να το πούμε όμως προς τα έξω και εμείς και εσείς όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία και αυτό θα μπορέσει να αλλάξει τις πολιτικές. Τέλος, δύο-τρία λόγια για τη διεθνή συνεργασία. Προφανώς αυτό είναι κάτι που χρειάζεται παντού. Οι πλούσιες χώρες έχουν μια ειδική ευθύνη ιστορική λόγω των σημερινών επιπέδων εκπομπών, λόγω της πρόσβασης στη τεχνολογία και μπορούν να δώσουν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να δείξουν με το παράδειγμα ότι αυτή είναι η διέξοδος από την ύφεση. Τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει, υπάρχει πολύ ρευστό στη κοινωνία μας. Υπάρχουν ε, πόροι που δεν χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η στιγμή τώρα για να ορίσουμε τη βάση για μακροπρόθεσμη σοβαρή ανάπτυξη. Όχι αυτές οι φυσαλίδες που είδαμε στο παρελθόν. Όχι, θα πρέπει να ε, θέσουμε τώρα τα θεμέλια για ισχυρή ανάπτυξη. Είναι κακό να δούμε την ύφεση σαν ένα λόγο δισταγμού. Όχι του αντίον, θα πρέπει να είμαστε τολμηροί. Θα πρέπει να μην περιμένουμε. Υπάρχει και κάτι θετικό. Εμείς διστάζαμε και ορισμένοι παρακολουθούσαν, αλλά σε ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Ιδονησία, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια είδαμε να κινούνται προς τα εμπρός. Οι περισσότεροι από εσάς βέβαια δεν διαβάζω κάθε βράδυ τα πενταετή προγράμματα της Κίνας. Εγώ θα σας έλεγα να διαβάσετε την ε, περίληψη του 12ου πενταετούς ε, προγράμματος που δημοσίευθηκε τον Οκτώβριο και θα δημοσιευθεί σε λεπτομέρειες ε, την Άνοιξη. Θα είμαι με άλλους ηγέτες τον Μάρτη σε ένα, σε ένα συνέδριο όπου θα καθοριστούν ορισμένοι κλάδοι που θα αυξηθούν από το 3% της οικονομίας στο 15% τα επόμενα 10 χρόνια. Καθαρές τεχνολογίες, ε, απολυσματική χρήση ενέργειας, ε, παραγωγή, τρένα υψηλής ταχύτητας παραδείγματος χάρη, βιοκαύσιμα, φύκια, ε, πληροφορική, κινούνται πάρα πολύ ισχυρά προς τις ε, βιομηχανίες που θα ηγηθούν της νέας αυτής ε, ε, βιομηχανικής επανάστασης. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν. Η Ανατολική Ασία ηγείται τώρα σιγά σιγά. Η Ευρώπη σιγά σιγά χάνει την ηγεσία που είχε, όπως είπε και ο πρόεδρος Περόζο. Εάν η Ευρώπη και η Κίνα ηγηθούν των θεμάτων αυτών θα μπορέσουμε να αναλάβουμε την ηγεσία των, σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν ήδη κινήσεις προ τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες εδώ για την Ευρώπη και έχει έρθει η στιγμή όχι για την τεχνοφροσύνη αλλά για να αλλάξουμε τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Να ατενίσουμε προς το μέλλον, να δούμε ποιε είναι οι νέες βιομηχανίες που θα ηγηθούν να ε, από αυτό που έχει γίνει και να διπλασιάσουμε τι προσπάθειές μας. Δεν είναι αυτή η στιγμή για δισταγμούς, αλλά για σαφείς ισχυρείς πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Λόρδε Στέρν, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή της συζήτησης και ότι είπατε ότι καινοτομία, τεχνολογίες, ε, ναύσματα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Χωρίς να μακρηγορήσω θα ήθελα αμέσως να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάρετ Φόρντ να μας παρουσιάσει την δική του άποψη. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να ευχαριστήσω και την αυτοεξοχότητα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα αστείο, να ρίξουμε φως στις σχέσεις μας με τους καταναλωτές γύρω από τον στόχο τον οποίο έχουμε. Τρία βασικά σημεία. Πρώτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω τα σημαντικά εμπόδια που βλέπουμε εμείς σαν εταιρεία Philips, ποια είναι τα εμπόδια, ποια είναι η αδράνεια που συναντάμε. Θα ήθελα να συζητήσω επίσης την αξιοπιστία κάποιων προτάσεων οι οποίες έχουν γίνει και τρίτον να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός για να προωθήσουμε τη σημερινή συζήτηση. Πρώτον, να πω ότι εμείς θεωρούμε ότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι το 50% του προβλήματος ή το 50% της δυνατότητας που έχουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ακριβώς ε, η κουλτούρα του χαμηλού εναρκτήριου σε εισαγωγικά κόστος. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζει ο καταναλωτής είναι το υψηλό κόστος. Αυτό δεν είναι θέμα καταναλωτή μόνο. Δεν είναι μόνο η συμπεριφορά του καταναλωτή εκεί που είναι τέτοια, αλλά και το δημόσιο και οι δημόσιες επενδύσεις ε, κοιτάνε ακριβώς την τιμή στην ετικέτα όλοι και όχι το μακροπρόθεσμο κόστος. Και αυτό έχει σαν συνέπεια την μεταφορά ουσιαστικά ε, του κόστου στις επόμενες γενναίες. Συνεπώς, εμείς πιστεύουμε ότι το πιο επίγον θέμα στην παρούσα κατάσταση είναι ακριβώς το θέμα της αντίληψης που επιβάλλει χαμηλό εναρτήριο κόστος. Το δεύτερο θέμα είναι το μέγεθος αυτής της ευκαιρίας που αντιμετωπίζουμε. Ακούσαμε από πάρα πολλούς συναδέλφους πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό και πώς μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία. Αλλά πάρουμε το φωτισμό. Το 40% του ηλεκτρισμού καταναλώνεται από το φωτισμό στην Ευρώπη. Αυτό μπορούμε να το μειώσουμε με τη σημερινή τεχνολογία κατά 45%. Καλό ακούγεται αυτό. Σε οικονομικό επίπεδο όμως σημαίνει 28 δις λιγότερο σε ετήσια βάση σημαντική μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα και αυτό φυσικά ε, μας δίνει τη δυνατότητα να μην δημιουργήσουμε 141 νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτά τα 300 δις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού λοιπόν. Βασικός μας στόχος λοιπόν είναι να συζητηθεί το θέμα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας πιο έντονα από ό,τι σήμερα. Αν έχουμε μια ενεργειακή αποτελεσματικότητα 1% το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι το 2050 ε, θα χρειαζόμαστε λιγότερους φυσικούς πόρους ε, κατά 140% καθαρούς πόρους βέβαια. Αν πάμε στο 3% θα χρειαστούμε το 40% των σημερινών ενεργειακών υποδομών να είναι καθαρές και αυτός ο στόχος νομίζω ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστος. Ταυτόχρονα πολλοί έχουν ήδη αναφερθεί στο ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρξει δράση, αν δεν υπάρξουν ξεκάθαροι στόχοι, που να στηρίζονται από ε, συγκεκριμένη παρουσία και ενέργειες. Και το τρίτο σημείο είναι αυτό στο οποίο δεν κοιτάμε πάρα πολύ συχνά και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πρίγκιπας της Ουαλίας. Όχι απλή καινοτομία, αλλά καινοτομία κατανοώντας ε, τα συμφέροντα των καταναλωτών. Μην υποτιμάμε την εξουσία που έχουν οι καταναλωτές. Δεν μιλάμε για την απλή λαϊκή εξουσία ή την εξουσία που έχει ο απλός πολίτης, αλλά βλέπουμε ότι πάρα πολλά θα έλεγα καθεστοτικά σημεία του τρόπου σκέψης των πολιτών πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Πρέπει να υπάρξουν επαναστάσεις σε εισαγωγικό όπως έχουν υπάρξει επαναστάσεις στον τομέα της κοινωνικής δικτύωσης σαν παράδειγμα. Η κατανόηση λοιπόν από πλευράς του πολίτη των θεμάτων που μας απασχολούν δεν θα πρέπει να είναι κάτι το, στο οποίο θα καταλήξουμε σαν συνδυασμός ή να είναι ταυτόχρονα κάτι το οποίο θα είναι αυστηρά διασκεδαστικό και ευχάριστο. Όχι. Εγώ νομίζω ότι αν μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο ευχάριστο και στο δυσάρεστο, αυτό που ονομάζουμε σαν παράδειγμα δυναμικός φωτισμός, μπορούμε εμείς να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας από ένα σχολείο κατά 40%. Αυτό δεν προκάλεσε καμιά ιδιαίτερη προσοχή, αλλά ταυτόχρονα κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις στον τομέα του, του χρωματισμού του φωτισμού, μπορέσαμε να αυξήσουμε την ταχύτητα ανάγνωσης των παιδιών κατά 30%, μειώσαμε την ανορθογραφία των παιδιών κατά 40% και μειώσαμε και τις απουσίες κατά 70%. Ποιος γονιός δεν θα μπορούσε λοιπόν να πιστεί από τους στόχους αυτούς που είναι φυσικά η εκπαίδευση των παιδιών μας αλλά στην περίπτωση που μιλήσουμε μόνο για την ενέργεια και αυστηρά για την ενέργεια το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δεύτερον, τι λόγο χρησιμοποιούμε. Όταν μιλάμε για δυναμικό φωτισμό δεν λέει πολλά πράγματα. Όταν μιλάμε για ενεργειακή αποτελεσματικότητα πολύ βαριούνται. Όταν μιλάμε για πρασίνισμα είναι πολιτική επιλογή. Εμείς προκαλέσαμε λοιπόν το ενδιαφέρον και των γονιών και των παιδιών και των ε, φυσικά διδασκόντων. Θα πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν μια εικόνα μια ζωή η οποία είναι καλύτερη από τη σημερινή, δεν απειλείται και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του καθημερινού ανθρώπου. Η συζήτηση μέχρι τώρα ήταν δεοντολογική, περιβαλλοντική, πολιτική, οικονομική αλλά αυτό δεν φτάνει. Αν δεν αλλάξει τη συμπεριφορά του ο πολίτης σε καθημερινή βάση δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος με τον πολίτη και να υπάρξει αυτή η επανάσταση την οποία όσοι όλοι εμείς επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος, Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, εμεί είμαστε υποφασιστικοί για το μέλλον διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Θα πρέπει οι ελπίδε μα να μεταφραστούν σε πράξει, να πραγματοποιήσουμε το όραμα το οποίο έχουν κατά νου οι ηγέτε Ευρώπη. Πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα σήμερα και να καλυφθούν από οικονομική υποστήριξη. Χαιρόμαστε για την ισχυρή εταιρική σχέση που δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα μηδέν μηδενικών εκπομπών, αλλά μόλις ξεκινήσαμε. Ο καθίστον είπε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ αφενός και είπα και, και Κίνα και Ινδία αφετέρου, ότι οι μεν υστερούν, ή δε προχωρούν. Αυτό βέβαια σχετίζεται ε, και με τον τρόπο με τον οποίο έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σκέψεις σωστού αντιτίμου για τα χρήματα γιατί τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν σημαντικά ε, οικονομικά προβλήματα. Θα πρέπει μια προσέγγιση της σωστής αξίας για τα χρήματα για το διοξείο του άνθρακα σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε το σχήμα στο να κάνουμε αυτό που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Ποιοι είναι οι δύο τομεί που θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό ε, Ίδρυμα για το Κλίμα και το χρονοδιάγραμμά του σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της, ε, του περιορισμού του διοξιδίου του άνθρακα και της ε, ευημερίας Για τις περισσότερες χώρες ε, η, η ανάπτυξη ε, φυσικού αερίου σαν πρώτη πηγή ε, ενέργειας θα μειώσει τα διοξίδια του άνθρακα, το διοξίδιο του άνθρακα και θα οδηγήσει και σε άλλα ωφέλη, όχι μόνο την τήρηση των προτύπων. Ίσως γνωρίζετε μια έκθεση McKenzie που λέει ότι η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου θα προστατεύσει εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και θα μειώσει και το κόστος ενέργειας και ταυτόχρονα θα ε, πετύχει τους στόχους για το 2015. Λοιπόν, προώθηση του φυσικού αερίου θα μπορέσει να αυξήσει την υποστήριξη του κοινού, της κοινή γνώμης για τις απαραίτητες αλλαγές. Επίσης, Χρειάζεται να προωθήθει η προστασία, η συλλογή του, του άνθρακα. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη σχετική νομοθεσία, αλλά δεν ξέρω γιατί χρειάζεται να περάσουν δύο χρόνια μέχρι χρηματοδότηση είναι δυνατή. Η βιομηχανική κλή είναι έτοιμη να προωθήσουν το CCS. Αυτό είναι όμως δυνατό μόνο εάν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε γλίγορα τα ε, πιλωτικά προγράμματα. Επίσης θα πρέπει να δοθεί η συγκεκριμένη όθηση στην ενεργειακή αποτελεσματική χρήση ενέργειας το σωστό να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα με το 2030. Ένα παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασιλείο η Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος προτείνει για το 2030 να μειώσει τους στόχους της κατά 60% από τα επίπεδα του 1900. Αυτό σημαίνει μηδενικές εκπομπές από την παραγωγή ενέργειας μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει σημαντική αλλαγή από τη σημερινή κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει τεράστια επιτάχυνση των ε, σχετικών πολιτικών δράσεων. Το Ηνωμένο Βασίλειο τα σκέφτεται αυτά στα πλαίσια συμπληρωματικών ε, εγχώριων πολιτικών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι δημοκρατίας και ότι εκεί θα πρέπει να δράσουμε. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κομισιόν ε, πριν από λίγο έκλεισε τα κύρια στοιχεία της ε, τρίτης φάσης του ε, σχεδίου ανταλλαγής πιστοποιητικών εκπομπών. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα τόσο χρόνια για να περάσουμε στην τέταρτη φάση, γιατί θα πρέπει να είναι γνωστό το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις επενδύσεις μας. Φέτος θα πρέπει να εξετάσουμε την φάση 4 και του χρόνου να περάσει αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει οι βιομηχανικοί κύκλοι να γνωρίζουν ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό. Θα πρέπει να διεξασφαλίσουμε κύριε Πρόεδρε οι, γρήγο, οι πιο γρήγορε και οι πιο φτηνές ε, τεχνολογίες να μπορέσουν να προωθηθούν το γρηγορότερο δυνατόν και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη μας σε μέσα όπως το EDS για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας και να προχωρήσουμε προς μια ε, οικονομία χαμηλών εκπομπών. Το ρολόι προχωράει πρόοδε, δεν μπορούμε παρά να πετύχουμε πρόοδο από κοινού και προσβλέπω σε επικοδομητικό έτος με σωστή πρόοδο, με όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να έχουμε μια ευημαρία της Ευρώπης που να χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η συνάλφος Τίκαο είναι η πρώτη που θα μιλήσει αυτή τη στιγμή. Έχει τότε να κάνει μια σύντομη εισαγωγή και μια ε, σύντομη παρέμβαση. Παρακαλώ. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Transportul este coloana vertebrală a οι μεταφορές. Είναι στην ουσία η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ταυτόχρονα οι μεταφορές θα πρέπει ε, να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους ε, στη μείωση των εκπομπών και να πετύχει ε, το στόχο της Ευρωπαϊκή Ένωση της μείωσης δηλαδή του 20% των εκπομπών μέχρι το 2020. Είδαμε τι λέγει η Λευκή Βίβλος ε, για το μέλλον των μεταφόρων στην Ευρώπη. Μάλλον το κείμενο αυτό θα δημοσιευτεί στην τελική του μορφή τον μήνα Μάρτιο. Και σε επίπεδο συντονιστών βέβαια είχαμε προκαταρκτικές συζητήσεις με τον Επίτροπο Σιμ για να δούμε ποιοι θα είναι οι βασικοί στόχοι για τις βαθιές αλλαγές που θα πρέπει να υποστούν οι μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προβλήματα όπως η δυσκολία της κυκλοφορίας της πόλης, η μείωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων μεταφορέων, εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αυτών. Όλα αυτά είναι σημαντικά προβλήματα και πρέπει να οδηγηθούμε σε λιγότερη ανάγκη από τέτοιου είδου καύσιμα στις μεταφορές και θα πρέπει να διευκολύνουμε επίσης και τη ρευστότητα των συγκοινωνιών και φυσικά και το κόστος των φαινομένων αυτών στο περιβάλλον. Θυμίζω ότι 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ απορροφάται ουσιαστικά από την, απορροφάται για την αντιμετώπιση των συνοπιών της δυσκολίας της επικοινωνίας, ιδιαίτερα τις οδικές. Και το κόστος της υποδομές είναι πάρα πολύ δυσβάστακτο. Οι υποδομές στις μεταφορές δεν αναπτύσσονται με το σωστό τρόπο στην Ευρώπη. Δεν εφαρμόζονται σωστά τα προγράμματα και υπάρχει ουσιαστική ε, έλλειψη ε, σωστών καθορισμών προτεραιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει υπάρξει λοιπόν σημαντική πρόοδος όπως σαν παράδειγμα στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και δεν έχουν υπάρξει ε, σημαντικά βήματα προόδου, καθοριστικά βήματα προόδου και στον καθορισμό του ενιαίου συστήματος διαχείρισης του εναερίου χώρου. Πολλά μένει να γίνουν και εκεί και στον τομέα ε, επίσης ε, των εσωτερικών ε, υδάτινων μεταφορών. Απαιτείται παραποτάμιες μεταφορές κτλ. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξουν νέες προτάσεις και στον τομέα των πολυτροπικών μεταφορών, της δημιουργίας hubs, κέντρων δηλαδή συντονισμού των μεταφορών και απαιτείται να υπάρξουν και αλλαγέ στον τομέα των δημοσίων προμηθειών έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται πιο πράσινα οχήματα στις δημόσιες μεταφορές. Ταυτόχρονα η φορολογική πολιτική θα πρέπει να βοηθήσει ε, στο να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα την έρευνα και την ανάπτυξη για έξυπνα συστήματα μεταφορών και γενικότερα θα πρέπει να προωθήσουμε νέες αντιλήψεις και νέες συμπεριφορές στους πρωταγωνιστές των μεταφορών. Ακόμα και επιμέρους τομείς όπως η τιμολογιακή χρήση των υποδομών μεταφορών είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συντάξει μια έκθεση νέας ιδίας πρωτοβουλίας για τη Λευκή Βίβλο μόλις μας τη στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς στιγμή θα ήθελα να κάνω απλά μία αναφορά στη νέα στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη θα πρέπει επιτέλους να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο τους φυσικούς πόρους που έχει στη διάθεσή της. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε στο μεσοπρόθεσμο μέλλον το 2050 να μειώσουμε κατά 80 με 90% τις εκπομπές καυσαερίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο άπτεται άμεσα των μεταφορών φυσικά και συνολικότερα βέβαια του περιβάλλοντος. Περιμένουμε λοιπόν τις τελικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη, όπως επίσης και το στρατηγικό πρόγραμμα για την τεχνολογία γιατί οι μεταφορές περισσότερα από οτιδήποτε άλλο χρειάζονται από την καινοτομία ε, όπως επίσης ε, και ε, νέες μορφές επιστημονικής ρύθμισης των προβλημάτων τους. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να σας υποχρεώσω η συζήτηση να γίνει στο προηγούμενο χρόνο. Αδύνατον σχεδόν. Αλλά σας παρακαλώ, ας προσπαθήσουμε να έχουμε παρεμβάσεις του ενός λεπτού για να μπορέσουν και οι τρεις επισκέπτες μας να απαντήσουν. Η συνάδελφος Χάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Λόρδο Στέρν. Είσαστε ένας ε, πολύ γνωστός ε, οικονομολόγος και θα ήθελα να ξέρω ποια θα ήταν η ε, συμβουλή σας για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμα θέλουμε να ε, μειώσουμε τον εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα από το μείον 30 που τη στιγμή στο μείον 30 τι θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν συζητάνε αυτό το θέμα Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κλούτ μας. Μία ερώτηση προς τον κύριο Στέρν και προς τον κύριο σου είναι, η Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόσκληση ε, ευρωβουλευτών να είμαστε αντίθετοι από, από με, τα, με τα ε, standard, με τα benchmarks. Ποια είναι η δική σας ε, στάση αυτή η πρόσφατη απόφαση για το benchmarking, για το καθορισμό ποια είναι. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Φόρντ. Έχουμε απαγόρευση τους ανεπαρκείς ε, λαμπτήρες φωτισμού στην Ευρώπη. Αυτό θα επιταχύνει την καινοτομία. Πώς εξελίχθηκε δηλαδή η αγορά από τότε που το εισήγαμε αυτό το μέτρο. Πρώτα σας ευχαριστώ. Έντσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έχω μια ερώτηση για τον κύριο Hans van Αυτό είναι το, το όνομά σας, από ό,τι κατάλαβα. Της Shell. Από ό,τι κατάλαβα, η εταιρεία Shell έχει ένα 60% στο σχέδιο πετρελαίου στην Ακαμπάσκα. που από 70.000 ε, χιλιάδες βαρέλια ανά ημέρα, τώρα προωθείται στα 150.000. Ποια είναι τα μέτρα που έχει κατά νου η ΣΕΛ για την αποθήκευση του άνθρακα για να μειώσει τις εκπομπές διοξίου του άνθρακα από, τις, από τα κοιτάσματα αυτά. Πρώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει κανένα άλλο ζητήσει το λόγο. Δεν θα δώσω το λόγο στους κυρίους εδώ. Θα αρχίσω με τον Λόρδο Στέρνα. Uh, uh, για την κυρία Χάση. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα για να περάσουμε από το 20% στο 30% είναι ε, ηχηρά. Υπάρχουν τρία θέματα όμως τα οποία πρέπει να υπογραμμίσουμε. Πρώτον, από τη μία επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον, αλλά αυτό θα το πετύχουμε με ρευστότητα από τη μία και λιγότερη πίεση στους φυσικούς πόρους από την άλλη. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δεύτερον, η ιστορία των βιομηχανικών επαναστάσεων δείχνουν ότι οι επενδυτικές ροές πηγαίνουν στους πρωτοπόρους και στην περίπτωση αυτή οι πρωτοπόροι θα είναι αυτοί που θα σκεφτούν το μέλλον και θα εφαρμόσουν σωστά την πολιτική τους. Και τρίτο, έχουμε ένα πολύ ισχυρό διεθνές μήνυμα. Οι πλούσιες χώρες φάνηκε ότι διστάζουν, ενώ κάποιες άλλες προχωρούν γρήγορα. Συνεπώς εδώ βλέπουμε ότι και οι δύο κατευθύνσεις, και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω, υπάρχει αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη. Όλες οι χώρες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό διευκολύνει τις διεθνείς συμφωνίες. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ναι μεν έχουμε την οικονομική κρίση αλλά και για αυτά τα οποία είπα και για τα μηνύματα στα οποία αναφέρθηκα θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να περάσουμε στο 30% γρήγορα. Δεύτερον, για τα λεγόμενα benchmarks. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμείνει στις φιλοδοξίες της. Η ιστορία μας δείχνει ότι κάθε φορά που εξετάζει κανείς το κόστος σαν παράδειγμα των καταλυτών των αυτοκινήτων ή το κόστος ε, της ε, αμόλυβδης βενζίνης. Πάντα οι προβλέψεις ήταν καταστροφικές σε σχέση με το πιθανό τους κόστος. Αλλά αν πράγματι ξεκαθαριστούν οι συνθήκες και είμαστε πιστικοί, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να δει κανεί ότι η εμπιστοσύνη στις οικονομίες κλίμακας οι οποίες δημιουργούνται θα οδηγήσει σε λιγότερες ανησυχίες και σε ένα κόστος χαμηλότερο από το υποστηριζόμενο από τη βιομηχανία παλαιότερα. Ταυτόχρονα, αν κρατήσουμε την ηγετική θέση την οποία θέλουμε μέσω μιας ισχυρής Ευρώπης και σε συνεργασία με άλλα μέρη του κόσμου βέβαια, τότε οι κίνδυνοι των ενεργειών μας θα είναι πολύ μικρότεροι. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία μπροστά μας. Το κόστος είναι χαμηλότερο από ό,τι προβλέπετε και έχουμε και την δυνατότητα σε αυτή τη φάση της διεθνούς συνεργασίας Όλα αυτά είναι επιχειρήματα έτσι ώστε να εμείνουμε στους στόχους μας. Δεν είναι καιρός για δισταγμούς και για δηλία. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Ευχαριστώ πολύ, κ. Um, um, Ευχαριστώ για την ερώτηση Κλοντ για τα benchmarking. Γνωρίζω τη συζήτηση η οποία γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αν εφαρμόσετε κάποια τέτοια benchmarks σε τομείς που καλύπτονται από τα ETS, τότε στην ουσία υπάρχει μια νομική επικάλυψη. Αλλά αν επιβάλλετε δύο μορφές νομοθετικής ρύθμισης, τότε αγνοούμε τα πλεονεκτήματα των ETS, γιατί στην ουσία το ETS είναι ένας πίνακας βαθμολογίας της χαμηλότερης παραγωγής διοξίδιου του άνθρακα σε επίπεδο οικονομικό, δηλαδή σε επίπεδο κόστους, είναι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε με τον ευθυνότερο δυνατό τρόπο πρώτα τις εκπομπές καυσαερίου. Ερώτηση Χούσκη σχετικά με τα ταμπάσκα. Δεν ξέρω ακριβώς αν μιλάμε για το 60% αλλά είμαστε μέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια εκμετάλλευσης. Έχει διευρυνθεί τελευταία. Τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε μειώσει την παραγωγή συνθετικού πετρελαίου κατά 40% τα τελευταία 25 χρόνια. 40%. Σε αυτή τη φάση γενικά έχουμε προχωρήσει να μειώνουμε πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη παραγωγή πετρελαίου στην Βόρεια Αμερική. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της μείωσης δηλαδή, ιδιαίτερα σε σχέση με το CTS και με τη βοήθεια της κυβέρνησης της πολιτείας της Αλμπέρτα η οποία επενδύει ε, πολλά εκατομμύρια καναδικά δολάρια στο πρόγραμμα Quest. Και γι' αυτό η παραγωγή ε, πετρελαίου από αμμώδεις ασφαλτούχες περιοχές είναι το κόστος χαμηλότερο από την εξόριξη την παραδοσιακή σε άλλες περιοχές της Βορειοαμερικής. Στην Αλμπέρτα Έχουμε να κάνουμε με φυσικούς πόρους οι οποίοι δεν έχουν ανάλογο τους στον κόσμο εκτός από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό λέγει πολλά. Δεν είναι μεγάλο δώρο λοιπόν να έχουμε αυτή τη στιγμή ε, τόσο τεράστιους πόρους που να μην ελέγχονται από χώρες του ΟΠΕΚ. Πρέπει λοιπόν μέσω της καινοτομίας να μετατρέψουμε τους πόρους αυτούς σε αηφόρους πόρους και πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις καναδικές αμμώδεις ασφαλτούχες ζώνες και σε άλλες περιοχές τις οποίες υπάρχουν εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και μπορούμε να ανησυχούμε εκεί. Η απάντησή σας είναι ναι λοιπόν, αλλά να πω ότι το 2008 Στη Philips ε, υπήρχαμε πάρα πολύ ε, μικρό ποσοστό αυτών των νέων λαμπτήρων. Ε, στα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί το ποσοστό αυτό. Δεν είναι απλά εμπορική η επιτυχία μας. Είναι ότι ήμασταν αρκετά τολμηροί στο να επενδύσουμε εκεί που έπρεπε. Το ποσοστό που δίνουμε εμείς στην έρευνα και στην ανάπτυξη για, τους νέες, ε, για τις νέες μορφές φωτισμού είναι σχεδόν το σύνολο των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο. Η επιτάχυνση των διαδικασιών που ακολουθούμε ήδη είναι απαραίτητη και υπάρχει δυνατότητα για βιομηχανικές χρήσεις σαν παράδειγμα να υπολογίζεται το κόστος απόλυτα. Ο απλός καταναλωτής βέβαια δυσκολεύεται στο να κατανοήσει, περνάει από ένα παραδοσιακό λαμπτήρα θέρμανσης σε έναν λαμπτήρα νέου τύπου, βλέπει μόνο τη διαφορά στην τιμή σε μια πρώτη φάση. Τώρα όμως σιγά σιγά κατανοεί ο πολίτης ότι και λόγω της τιμής και λόγω των προβλημάτων που έχει η εσωτερική αγορά πλημμυρίστηκε, ε, πλημμύρισε συγγνώμη, η εσωτερική αγορά από προϊόντα χαμηλής ποιότητας και αυτό δημιούργησε μια κάποια απογοήτευση ε, στο στον πολίτη. Λοιπόν, έχουμε πείσει του επαγγελματίε χρήστε. δεν έχουμε απόλυτα πείσει του μεμονωμένου καταναλωτέ πολίτε, αλλά παρόλα αυτά ε, ε, διευρύνουμε συνεχώ την κάμα των προϊόντων μα και η πορεία που κάναμε μέχρι τώρα, που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα ήταν η σωστή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Το πρόβλημα αυτών των συζητήσεων είναι ότι υπάρχει κίνδυνο να παρεμβαίνει κανένα πολύ στα γενικά. Δεν έχουμε χρόνο. Τα προβλήματα βέβαια είναι στις λεπτομέρειες. Θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μάλκον Χάρμπορ που προεδρεύει το επόμενο πάνελ. και κύριοι, θα έρθουν σε λίγο οι εμπειρογνώμονες εδώ για να ξεκινήσουμε το τελευταίο πάνελ. So a very uh, welcome from, uh, me, uh, Malcolm θα ήθελα να σα καλωσορίσω. Εγώ είμαι Μαύρο Χαμπέρ, είμαι τη τη Επιτροπή Ιστορικής Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πάρα πολύ ελκυστική αυτή η ημέρα σήμερα και θα συνεχίσω την τόσο σημαντική συζήτηση πάνω στο βασικό θέμα μείωση του άνθρακα στην ε, βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα. Όπως ελέγχθη προηγουμένως, μέσα στα πλαίσια του γεγονότος ότι την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, ιδίως στις ε, διεθνές αγορές, θα πρέπει να ε, την προσέγγιση μας και βέβαια η προσέγγιση της μείωσης του άνθρακα ε, θα είναι πάρα πολύ ουσιαστική για την βιομηχανία και για την παραγωγή ενέργειας. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντες εμπεριγνώμενες εδώ και ελπίζω να έχουμε και κάποιο χρόνο γιατί έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές εδώ. Ο κύριος μας ομιλητής είναι ο Δόκτωρ Ότμαρ Έτενχόφερ, που είναι συμπρόεδρος ε, του Σωμάτας Εργασίας 3 για την αλλαγή του κλίματος και είναι επίσης ε, αντιπρόεδρος και κύριος οικονομολόγος του Ινστιτούτου για επιπτώσεις του κλίματος της έρευνας για το κλίμα στο Πότστον. Νομίζω ότι αυτή είναι εκείνη που προτιμά να συμβουλεύεται η Άγγελα Μέρκελ στο Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο Βερολίνου για Τεχνολογία. Έχουμε τον Φίλιπ Τελπέσ, πρόεδρο της ε, Carrier, γνωστή βιομηχανία για προϊόντα θέρμανσης και ψήξης που θα μας αναφέρει την αλλαγή της δικής του επιχείρησης. Μετά θα έχουμε τον Jules Gottenhaus, που είναι πρόεδρος μιας ε, επιχείρησης ε, πράσινης ενεργειάς της Topel Energy και κυρίως είναι ο κύριος διευθυντής ε, του, Ιδρυματο, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τις αλλαγές του κλίματος. Φιλανθρωπικό Ίδρυμα που δεν ε, έχει ούτε ιδεολογική ούτε πολιτική θέση. Λοιπόν, και τελευταίος αλλά οπωσδήποτε εξίσου σημαντικός είναι ο Λόιβα Σόρενσεν που είναι πρόεδρος της θεσμικής ομάδας επενδύσεων για τις κλιματικές αλλαγές. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι μας ε, έχουμε σημαντική ε, αρχή στις επενδύσεις για τις κλιματικές αλλαγές. Ε, η ομάδα αυτή έχει 65 μέλη, μεταξύ των οποίων και τα πιο μεγάλα ταμεία συνταξιοδότησης. Λοιπόν, αυτοί θα είναι οι κύριοι μας και μετά Ελπίζω να περάσουμε σε μια συζήτηση και θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ τον συνάδελφο Τζιλ Τσίτσεστερ που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Νοτιοδυτικό Αντιπρόκειο και ότι είναι μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας Ερεύνα και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το άλλο που θέλω να πω και σημείωσα κάτι που είπε ο, προ, ο πρίγκιπας της είναι cool να χρησιμοποιεί κανένα λιγότερο και εμείς τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ε, προηγμένη τεχνολογία, ένα ρολόι έχω εδώ 10 λεπτά για τον δόκτωρα Οντενφέ, 5 λεπτά για τους άλλους πανελίστ και 3 λεπτά για τον Τζαλ Τσίσεστερ. Το ρολόι τρέχει. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ο Πρόεδρος ήδη αναφέρθηκε στα όργανα στα οποία εργάζομαι και είμαι και αντιπρόεδρος του IPCC και προσπαθώ να είμαι πάντα ιδιαίτερα αντικειμενικός. Τα επόμενα δέκα λεπτά όμως δεν θα μιλήσω σαν εκπρόσωπος του IPCC, και δεν θα σχολιάσω τις θέσεις του IPCC, αλλά αυτά τα οποία θα πω αφορούν εμένα προσωπικά και το Ινστιτούτο του Πότσταμ. Η πρώτη δήλωσή μου είναι σαφής. Αν συνεχίσουν τα πράγματα όπως είναι σήμερα δεν πάμε πουθενά. Οι περισσότεροι κλιματολόγοι πιστεύουν ότι το να αποφύγουμε τις επικίνδυνες κλιματολογικές αλλαγές πρέπει να μειώσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 με 2 βαθμούς. Αυτό θα κοστίσει κατά 1 με 2% του συνολικού ΑΕΠ μέχρι το 2050. Όμως, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω, η δυνατότητα που έχουμε είναι μικρή και μικραίνει συνεχώς. Αν συνεχίζουμε να επενδύουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι το 2030, το δύο, οι δύο βαθμοί που θα είχαμε σαν στόχο δεν θα είναι κάτι το εφικτό το να αναλάβουμε εμείς την λήψη αποφάσεων μέχρι το 2020 θα αυξήσουμε το κόστος αποκατάστασης κατά 50% ενώ κόστος αποκατάστασης, το κόστος αποκατάστασης των συνεπειών και των βλαβών από τις κλιματολογικές αλλαγές. Όλα αυτά λοιπόν τα κόστη αυξάνονται όσο υπάρχει αδράνεια από πλευράς μας. Νομίζω ότι ο πιο σημαντικός κίνδυνος για μια φιλόδοξη κλιματολογική πολιτική είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και η μείωση της τιμής του άνθρακα ή οι χαμηλές τιμές του άνθρακα. Η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας και το IPCC πιστεύει ότι ε, θα αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου τις επόμενες δεκαετίες ακόμα και αν εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία η οποία να λέει κάτι το διαφορετικό θα έχουμε τρεις συνέπειες από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ο άνθρακας θα γίνει πιο ανταγωνιστικό στην Ινδία και την Κίνα. Είδαμε ότι η εντατική χρήση του άνθρακα έχει αυξηθεί αντί να μειωθεί στους τομείς αυτούς και στις χώρες αυτές. Η εξόριξη μη παραδοσιακού πετρελαίου, επισυμβατικού πετρελαίου θα αυξηθεί από το 2011 μέχρι το 2035. Η Κίνα, η Ινδία θα επενδύσουν σε τέτοιου είδους μορφές ενέργειας και αυτό θα οδηγήσει σε μια παραγωγή ενός εκατομμυρίου ε, βαρελιών πετρελαίου επιπλέον το 2050. Η διαδικασία αυτή δεν θα σταματήσει από την έλλειψη Πορον άνθρακα. Ο άνθρακας είναι άφθονος, είναι πολύ φθηνός και δεν υπάρχει έλλειψη ορυκτών καυσίμων για τον υπόλοιπο του αιώνα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν υψηλέ τιμές του πετρελαίου και χαμηλές τιμές του άνθρακα είναι συνδυαστικά ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για την πολιτική στον τομέα του κλίματος. Αν τα μέσα τα οποία μας δίνει η ατμόσφαιρα στη διάθεσή μας είναι λίγα, τότε ένας τρόπος μόνο υπάρχει για να βγούμε από το δίλημα αυτό. Η τεχνολογία και η καινοτομία. Θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις δύο, αυτούς τους δύο παράγοντες για την πράσινη ανάπτυξη τότε θα μιλήσουμε για σωστούς τρόπους και οικονομικούς τρόπους αποκατάστασης των κλιματολογικών βλαβών. Η καινοτομία φυσικά είναι το κλειδί για την πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά δείχνουν ότι η απανθρακοποίηση σε εισαγωγικά απαιτεί να εντοπίσουμε σωστά τον στόχο της ανταγωνιστικότητα της ενέργειας σαν ένα στόχο ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραγνωριστεί. Κάποιες από τις τεχνολογίες βέβαια είναι πιο σημαντικές από άλλες. Εδώ καταρχάς το κόστος αυξάνεται βέβαια. Η ε, διαθεσιμότητα των μεθόδων αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα και εκμετάλλευσης αυτών των αποθηκευμένων ποσοτήτων ε, είναι κάτι το οποίο θα προσθέσει στο κόστος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αν δεν πάρουμε γρήγορα μέτρα το κόστος της αποκατάστασης μπορεί να διπλασιαστεί και δεν, μπορούμε να πετύχουμε τους, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε. Το ίδιο ισχύει επίσης και με τη χρήση της βιομάζας το κόστος της αποκατάστασης θα διπλασιαστεί μέσω της χρήσης της βιομάζας. Η βιομάζα είναι πολύ σημαντική βέβαια σε συνδυασμό με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα γιατί αυτό θα επιτρέψει την απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να δούμε ακριβώς κάπως και τι επιπτώσεις θα έχει στο κόστος το θέμα της αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων πράσινη ανάπτυξη λοιπόν απαιτεί ένα σταθερό δίκτυο το οποίο να είναι απεξαρτημένο από τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας. Αυτό χρειάζεται η Ευρώπη, αυτό χρειάζεται και περαιτέρω έρευνα και κίνητρα στον τομέα της αποθήκευσης του άνθρακα και ενίσχυσης φυσικά της παραγωγής ενέργειας και της προμήθειας ενέργειας από εναλλακτικές πηγές θα πρέπει να υπάρξει αποσύζευξη της οικονομικής ανάκαμψης από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και οι νέες επενδύσεις οι φιλικές για το περιβάλλον ε, θα είναι συμβατές με την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε ε, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί και από μια λογική τιμή του άνθρακα σαν πηγή ενέργειας. Μόνο η τεχνολογία θα πρέπει να επιβαρύνει βέβαια το κόστος του άνθρακα στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της πρακτικής και μέσω της έρευνας. Μια σωστή και αξιόλογη πολιτική στον τομέα της τιμολόγησης του άνθρακα θα πρέπει να συνοδεύεται και από την καινοτομία μπορεί η προσπάθεια αυτή να συμπληρώσει το, την επιρροή που έχει το κόστος του άνθρακα στις κλιματολογικές αλλαγές. Έτσι θα πετύχουμε τους στόχους μας με αποτελεσματικό τρόπο. Μια τεχνολογική πολιτική χωρίς έλεγχο της τιμής του άνθρακα τότε θα επιβαρύνει το κόστος της πολιτικής αποκατάστασης ε, σημαντικά. Να υπογραμμίσω εδώ κάτι το οποίο υπογράμμισε και ο Λόρδο Στέρν, απαντώντας σε μία από τις ερωτήσεις. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των κλιματολογικών εκ των κάτω προς τα πάνω και εκ των άνω προς τα κάτω. Είναι συμπληρωματικές αυτές οι δύο α, μέθοδοι. Βέβαια η Σύνοδος της Κοπενχάγης υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στη μέθοδο εκ των άνω προς τα κάτω από τις κυβερνήσεις και τις διεθνείς αρχές δηλαδή προς τη βάση. Παρ' όλα αυτά παραμένει απαραίτητο να συντονίσουμε τις πολιτικές μας και θα πρέπει οι εσωτερικές πολιτικές σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο περιφερειακό να ελέγχουν τις ε, προσπάθειες που γίνονται για τη μείωση του κόστους της ενέργειας και να συνδυαστούν για να είμαστε φιλόδοξοι ε, <clears throat> στο μέλλον. Ε, σαν παράδειγμα η διάχυση διοξιδίου του άνθρακα ή από αποθηκευμένες πηγές είναι μια ανησυχία για το μέλλον. Αλλά νομίζω ότι μόνο λίγοι τομείς θα φυγούν, θα έλεγα, ε, συνολικότερα. Το θέμα είναι όταν η διαφυγή ε, διοξιδίου του άνθρακα με τέτοιο τρόπο επηρεάσει την τιμή της ενέργειας και έτσι υπονομεύσει την πορεία προς την πράσινη ανάπτυξη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη. Αρκετές περιοχές του κόσμου αντιμετωπίζουν σοβαρά μια πολιτική ουσιαστική στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος το 25 ετές πρόγραμμα της Κίνας έγινε αντικείμενο αναφοράς από τον Λόδο Στέρν. Το θέμα των μελλοντικών περαιτέρω μειώσεων των εκπομπών είναι κάτι το οποίο θα θέσει το πρόβλημα του συνολικού κόστου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μείωση κατά 30% μέχρι το 2020 είναι ένας αξιόπιστος στόχος για το πέρασμα σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, σε μια σταθεροποίηση των επενδύσεων για την καινοτομία και για σωστούς στόχους για μετά το 2020 έτσι ώστε να φτάσουμε στο 2050 στο 80 με 90% μείωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα ενδιάμεσα μέτρα στη δεκαετία, σε 30 και σε 40 χρόνια από σήμερα. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι από θεσμικής πλευράς ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της, α, α, της πράσινης ανάπτυξης είναι το νέο ETS πρέπει να είναι σφαιρικό, συνολικό, να συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς των αυτό ETS και μέσω του συστήματος ανταλλαγής ποσοτήτων και θα επηρεάσει και τον καθορισμό των τιμών της ενέργειας. Νομίζω ότι το EU ETS έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία για μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σαφής ε, και πλούσια η παρέμβασή σας. Περνάμε στον Φίλιπ Τελπέσιο. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα πω ποιε είναι απόψει βάσει των εμπειριών που έχω από την αγορά και ορισμένα πρακτικά αποτελέσματα, ε, παραδείγματα για να δείξω ότι θα πρέπει να εργαστούμε σωστά προ σωστή κατεύθυνση. Στην, ε, εργάζομαι στην Ασία, Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, δεν βλέπω να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Η συνεργασία μας βασίζεται στην ε, αεροφυγική και στις τεχνολογίες για κτίρια και βάσω αυτή στα τα παραδείγματά μου. Έχουμε 70.000 ε, απασχολούμενους στην κατασκευή κτίριων Και τι γίνεται στι ε, διεθνεί αυτές ε, εταιρείε. Ε, επενδύουμε στην έρευνα και στην άπτυξη, στην παραγωγή, σε εκείνο το τομέα του κόσμου που κινείται πρώτος όσον αφορά την νομοθεσία. Αν έχετε μια νομοθεσία που είναι πιο καινοτόμη και πιο αυστηρή, η τοπική έρευνα και ανάπτυξη αρχίζει να βασίζεται πάνω σε αυτά και εξάγει μετά τα αποτελέσματα της έρευνάς Είμαστε οι πιο προηγμένοι εταιρείε αυτά στην Ευρώπη και θα σα δώσω ορισμένα παραδείγματα, σα δείξω ότι είναι δυνατό σε ορισμένες χώρες. Ε, το ένα παράδειγμα σχετίζεται με την ασφάλεια της τροφιμικής αλυσίδας. Τα περισσότερα τρόφιμα που πάνε στις αστικές περιοχές είναι ή κατεψυγμένα ή φρέσκα. Σήμερα χρησιμοποιείται ένα αέριο το οποίο κρατάει τα τρόφιμα φρέσκα μέχρι να φτάσουν στο σούπερ μάρκετ. Σε, μια, ε, σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχει 1,7 τόμος ε, του αερίου αυτού το οποίο ε, κρατάει τα τρόφιμα φρέσκα. Το κόστος είναι πολύ σημαντικό κάθε χρόνο και αυτό δημιουργεί το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Από εκεί προέρχεται το διοξείδιο του άνθρακα. Όχι από την ενέργεια. Εάν χρησιμοποιηθεί αντί του αερίου αυτό διοξείδιο του άνθρακα, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί η παραγωγή αυτή τη στιγμή εκπομπές είναι όπως από 400 αυτοκίνητα το χρόνια. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ναι, γίνεται. Υπάρχει μια χώρα τα, το που το κάνει. Ναι, η Δανία δεν χρησιμοποιεί αυτό το αέριο εδώ και πολλά χρόνια και τα τρόφιμα είναι εξίσου φρέσκα και φτηνά στην Δανία όπως και αλλού. Άλλες χώρες, Νορβηγία, Ελβετία, λίγες χώρες μέλη όμως. Μπορούμε να προχωρήσουμε γλίγορα, ναι. Αν το κάνουμε θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στην ε, ε, έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, στην παραγωγή στην Ευρώπη, στην υπηρεσία στην Ευρώπη και η ΕΠΑ και η Ασία θα έρθουν να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά στις τεχνολογίες μας. Χρειαζόμαστε χρήματα και ε, νόμους και ελέγχους. Δεύτερο παράδειγμα, από τα κτίρια. Ποιοι έρχονται εδώ όταν υπάρχει εξοπλισμός ενός μεγάλου κτίριου όπως αυτό οι τράπεζες. Η, η μηχανική. Ποιος πληρώνει το, το κόστος. Ο τελικός χρήστης, ο οποίος όμως δεν μπορεί να παρέμβει στις, για να γίνουν εξοικονομήσεις γιατί πολύ αργά φτάνει στη διαδικασία. Όλα παίζουν ένα ρόλο. Η ψήξη, του κτηρίου, η θέρμανση, τα παράθυρα, ε, τα, ο φωτισμός. Αλλά είπαμε, ο τελικός δεν προφταίνει να παρέμβει εκεί. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα για να γίνονται όλα στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη, ψήξη στα κτίρια στην ε, Ιαπωνία ε, είναι ε, εκεί που προηγούνται γιατί αναπτύχθηκε εδώ και 10 και 15 χρόνια. Ας πούμε το αντίθετο στη ΣΥΠΑ ήταν φτηνά τα καύσιμα και χάσανε τις αγορές και ε, δεν χρειάστηκε δηλαδή να προσπαθήσουν, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσουν οι τιμές ε, τους στο παγκόσμιο επίπεδο και τότε Χρειαζόμαστε λοιπόν στην Ευρώπη να έχουμε ενεργητικό ε, ρόλο, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε από εσά είναι η ταχύτητα, σαφή νομοθεσία, έλεγχη, όχι πάντα χρήματα, καμιά φορά ναι, γιατί ορισμένε τεχνολογίε χρειαζόνται μια βοήθεια για να ξεκινήσουν. Ιδίω στον τομέα τη αποτελεσματική χρήση τη ενέργεια δεν μπορεί να αυξηθεί δραματικά σε πολλού τομεί με τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σαφή και πάρα πολύ πρακτικά εφαρμόσιμα. Ο κ. Σκόρτμεγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Νομίζω ότι το επιχείρημα για το ποιο ρόλο πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακούστηκε από όλους σήμερα το απόγευμα και με πολύ πιστικό τρόπο. Μόνο αν κερδίσουμε θα έλεγα αυτήν την επόμενη βιομηχανική επανάσταση τότε θα σώσουμε τον πλανήτη αυτό και για τις επόμενες γενιές και απ' την άλλη να δημιουργήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης για τα παιδιά μας. Νομίζω ότι το δεύτερο μάθημα από αυτά που άκουσα σήμερα είναι ότι όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να βοηθούν τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης και όχι να τον παρεμποδίζουν. Και αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο έχουν πάρει οικονομολόγοι εδώ και αρκετό καιρό. Αν θέλετε να δώσετε κίνητρα στην εσωτερική σας βιομηχανία, θα πρέπει να διασφαλίσετε τον ανταγωνισμό και μια καλά ρυθμισμένη αγορά. Με χαρά άκουσα τον κύριο Φόρντι από τη Φίλιπς, να λέει πόσο σημαντικό είναι ε, το θέμα της νομικής ρύθμισης ε, της αγοράς λαμπτήρων. Οι παραδοσιακές οικονομικές αναλύσεις βέβαια δεν μας δείχνουν ακριβώς το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς αυτήν τη νέα οικονομική επανάσταση παραδοσιακά συστήματα εξισορρόπησης δεν συλλαμβάνουν το πλήρες εύρος της ε, ανατροπής που έχει συντελεστεί. Βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει με την βιομηχανία της πληροφορίας. Στα αυτοκίνητα τα οδηγεί κανείς πλέον μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ουσιαστικά. Και το ίδιο ισχύει επίσης και για τις οικοδομές και η διασταύρωση από τον ένα τομέα στον άλλον είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια, αλλά δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο ωφεληθούμε. Νομίζω ότι και επενδύσεις από άλλους τομείς, από δραστηριοποιούμενες σε άλλους τομείς επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ελκυστικό. Έχουμε λοιπόν εδώ τρεις τομείς τους οποίους πρέπει να εμείνουμε. Αν είσαι υπεύθυνο για μια επιχείρηση, έχει ένα όραμα για την επιχείρηση αυτό μακροπρόθεσμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αυτό. Λέει 80 με 90% μείωση το 2050. Έχετε θέσει ενδιάμεσα όμως και στους συγκεκριμένους απτούς στόχους για το 2020 και άκουσα και την αυτού εξοχότητα να λέει ξεκάθαρα σήμερα το απόγευμα ότι οι προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβονται το στόχους που θέτει η επιστήμη που είναι 30% και αυτό δεν είναι απαραίτητο μόνο για κλιματικούς λόγους. Είναι απαραίτητο γιατί πρέπει να λειτουργήσουμε ηγετικά στον συγκεκριμένο αυτό τομέα. Αν βάλουμε χαμηλούς στόχους, αν πούμε στους πληθυσμούς μας ότι εμείς δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί Οπότε ας μείνουμε στο 20% και ελπίζουμε να πάμε καλά μαζί με όλους τους άλλους. Αυτό δεν εμπνέει κανέναν. Αν έχουμε όμως φιλόδοξους στόχους και πούμε στους λαούς της Ευρώπης ότι εμείς θα ηγηθούμε τη επόμενης περιβαλλοντικής επανάστασης μέσω του στόχου 30% τότε δημιουργούμε τους στόχους που θα μετατρέψουν το όραμα σε πραγματικότητα. Ο επόμενος τομέας στον οποίο θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί είναι η αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας. Η τιμή βέβαια του άνθρακα από μόνη της δεν μα μας βοηθά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θα πρέπει να θέσουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους και για τους εξοπλισμούς τους ηλεκτρικούς και για τις κατασκευές και για την αυτοκίνητο βιομηχανία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε επίσης τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πάρουν νόμους που θα ανανεώσουν το χτισμένο μας περιβάλλον. Δεν πρέπει να περιμένουμε τον κύκλο των 40 χρόνων. Πρέπει να προχωρήσουμε σε καινοτομικά προγράμματα συντήρησης κτηρίων από τώρα. Και τώρα για το κλίμα. Έχει δημοσιευθεί ένας οδικός χάρτης για την περίοδο 2020-2050 είναι τεχνικά εφικτό να περάσουμε στην πλήρη απανθρακοποίηση σε εισαγωγικά μέχρι το 2050. Πρέπει να το κάνουμε αυτό και πρέπει να το κάνουμε μέσα σε μια ολοκληρωμένη κοινή αγορά, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφοράς ποσοτήτων και νομίζω ότι θα το κάνουμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Συνεπώς λοιπόν, εφόσον έχουμε ξεκάθαρους φιλόδοξους στόχους, εφόσον είμαστε αποτελεσματικοί και εφόσον εγκαταλείψουμε τον άνθρακα, τότε θα περάσουμε σε αυτήν την οικονομία της ευημερία και της έλλειψης υψηλών ποσοστών εκπομπών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για πάρα πολύ σαφή στοιχεία. Τέλος, ο κ. Σόρενσον. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε βουλευτέ, κύριε βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, η εισαγωγικά ότι τα είναι μια οργάνωση που οργανώνει τα, τους ε, ε Υπάρχουν και παρόμοια δίκτυα στην ε, Βόρεια Αμερική και στην Ασία. Πίσω μου βρίσκεται ο οποιοδήποτε μεγάλος ε, ε, θεσμικός επενδυτής ε, στην, ε, στον κόσμο και θα σας παρουσιάσω τις απόψεις τους. Λέμε ότι ένα από τα πιο ουσιαστικά πράγματα που θα πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια αν θέλουμε να καταπονομήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να περάσουμε σε ανάπτυξη είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρή και συνεχή διάλογο μεταξύ επενδυτών και νομοθετών. Γι' αυτό μια συνεδρίαση σαν αυτή τη σημερινή είναι πάρα πολύ καλό δεκτή από δική μας κοπιάς. σημαντικές επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν τα ε, επόμενη δεκαετία για να μπορέσουμε να περάσουμε στην ανάπτυξη με χαμηλή χρήση άνθρακα. 80% θα πρέπει να προέρχεται από ιδιωτικέ επενδύσει. Δηλαδή, οι ιδιώτε επενδυτέ έχουν ε, ουσιαστικότατο ρόλο να παίξουν στη μετάβαση στην οικονομία χαμηλής ε, άνθρακα. Η ικανότητά μα να παίξουμε τον ρόλο αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από την πολιτική. Ίσως αυτό δεν είναι η συνήθι ε, ε, ο συνήθις τίτλος, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι ισχυρή κυβέρνηση και περισσότερη νομοθεσία. Πάρα πολύ κυστικό. Χρειαζόμαστε πολιτικές που να μπορούν να υποστηρίξουν και να δεσμεύσουν τις επενδύσεις στην ε, ενέργεια με λίγο άνθρακα, αηφορία, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Χρειαζόμαστε ε, να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις κατά τη διάρκεια των ε, ε, επενδύσεων μας. Η πολιτική αυτή παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την διαφάνεια των επενδύσεων. Χωρίς τους επενδυτές δεν μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που θέλει να πάει ο κόσμος. Ελέγχθη ότι δεν υπάρχει έλλειψη κεφαλαίου. Πάντα υπάρχει κεφάλαιο. Αυτό ίσω που λείπει είναι η πολιτική βούληση να πληρώσουν για το κεφάλαιο αυτό ή να δώσουν το κατάλληλη προστασία για να ξεκινήσει να χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο αυτό. Κεφάλαιο υπάρχει πάντως. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές είναι αδιάφοροι κοινικά για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε των αντίον. Ανησυχούν πάρα πολύ οι περισσότεροι επενδυτές ανά τον κόσμο, αντιπροσωπίζουν τις κλιματικές αλλαγές, εξετίζουν στενά τις ευκαιρίες για τις κλιματικές αλλαγές και έχουν έντονη δεσμευσή για μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές που είναι σημαντικές για τις κλιματικές αλλαγές. Οι, οι θεσμικοί αυτοί οι επενδυτές δεν μπορούν να επενδύσουν ε, αν δεν είναι προς όφελος των πελατών τους. Όχι μόνο για κοινωνικούς λόγους, αλλά και για επιχειρησιακούς λόγους να προβλέπετε σημαντική εκκληστική επιστροφή. Αν δεν γίνει αυτό, οι επενδυτέ θα πάνε αλλού. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι επενδύσεις ε, γίνονται και εδώ και εκεί. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάρει τα χρήματα το πάει αλλού. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που είναι σημαντικό για τις κλιματικέ αλλαγές είναι ότι είναι κάτι που δεν είχαμε ούτε στην Κοπεχάγη, ούτε στην Κανκούν και ούτε στον Τάρμα που κατά πρόσωπο να το έχουμε. Θα πρέπει να παραμείνει ένας από τους κύριους στόχους για την πρόθεση της πολιτικής. Έτσι θα μπορούμε νομίζω να προχωρήσουμε πολύ πιο γλυκόρα. Από την άλλη μεριά, ε, διεθνής ε, συμφωνία δεν δίνει τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διακανονισμούς που χρειαζόμαστε για τη λήψη των αποφάσεων αυτών. Αυτό που χρειάζεται από την πολιτική είναι να δημιουργηθεί ίδιο ενδιαφέρον. Έτσι, να μπορέσουν αυτοί οι που διαχειρίζονται αυτά τα χαρατοφυλάκια να κάνουν αυτό που πρέπει. Δηλαδή, το να δοθεί η νομοθεσία αυτή σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε νομοθεσίε για την ενέργεια από τη δημιουργική χρήση ενέργεια, ε, ε, εκπομπέ αερίου του θερμοκηπίου κλπ. θα πρέπει να γίνουν ε, τα έξι. Καταρχήν, ε, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει πιο φιλόδοξου στόχου μέσω πρόθεσμα και όσον αφορά αποτελεσματική χρήση ενέργεια. Γιατί αν αποτυχούμε στον τομέα αυτόν, θα είναι το πιο ανώτο που μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερον, χρειαζόμαστε να υπάρχουν ε, πολύ φιλόδοξοι στόχοι για μακροπρόθεσμα. Μην ξεχνάτε ότι το 2020 για να επενδυτή είναι μεθαύριο. Τρίτον, θα πρέπει να δοθούν ε, τα σωστά κινήτρα από καλή και δημόσια πολιτική, συνεργασία διαμεθοριακά, η ε, υποστήριξη της ε, χρησιμοποίησης της ενέργειας, να μειωθούν οι επενδύσεις, οι επιδοτήσεις το γρηγορότερο δυνατόν και τέλος χρειάζεται οπωσδήποτε να δοθεί το εκ άνευ σταθερές και υψηλές τιμές, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε. Με δύο λόγια, αυτό θα χρειαστούν οι επενδυτές για να υποστηρίξουν ε, τις επενδύσεις τους. Στον τομέα αυτό και να προχωρήσουμε σε μια πράσινη οδό για να έχουμε τα σωστά ωφέλη από την ανάπτυξη, την ευημάρεια που μας υποσχέτει χρειάζεται η πράσινη πολιτική. Αυτό που χρειάζεται η πολιτική είναι να κάνει το σωστό χωρίς να κάνει το λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Μόλις ξεπεράσετε κατά λίγο τα πέντε λεπτά που είχατε στη διάθεσή σας. Πριν δώσω το λόγο στον Τσάλ Τσίτσιστα να πω ότι όποιος θέλει το λόγο μπορεί να τον ζητήσει. Δεν είναι αποκλειστική συζήτηση για ευρωβουλευτές και κάποιοι προσκεκλημένοι μας από άλλα όργανα μπορούν να ζητήσουν το λόγο. Κάποιοι από εσά έχετε ονόματα μπροστά σα, αλλά κάποιοι από το CLG σαν παράδειγμα μπορούμε το όνομά σας να σας δώσουμε το λόγο. Τσίτσεστερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να είναι ο τελευταίος είναι ότι έχουν φύγει τα μεγάλα ονόματα και μπορεί κανείς να είναι πιο χαλαρός και ανεπίσημος και να πει προκλητικά πράγματα. Δεν θα προσπαθήσω να κάνω κάτι τέτοιο βέβαια. Εγώ από το πρώτο μέρος της συζήτησης συγκράτησα κάποιες σκέψεις οι οποίες μου φαίνεται είναι άμεσα σχετιζόμενες με αυτά τα οποία ακούμε σήμερα. Καταρχάς, ο ρόλος του καταναλωτή. Νομίζω ότι ο καταναλωτής παίζει και κομβικό ρόλο. Και το να πείσουμε τον καταναλωτή να αλλάξει τις συνήθειες του είναι βασική πρόκληση. Ο Λόρδος Στέρν μας είπε ότι θα πρέπει εμείς να περάσουμε καλύτερα τα επιχείρηματά μας στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών. Είπε επίση ότι μιλάμε για μια βιομηχανική επανάσταση και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν επαναλάβει και άλλοι ομιλητέ. Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους μας. Και θα πρέπει να δούμε πώς οι προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις προχώρησαν. Τέθηκε ένα πρακτικό θέμα από τον κύριο Φόρντι της Φίλιπς, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της κουλτούρας του αρκτικού κόστους Πράγματι, σωστό είναι όμως και είναι να ανησυχεί ο κόσμος για την αρχική τιμή και πρέπει ακριβώς να πείσουμε τον πολιτικό κόσμο και τους βιομήχανους να ελέγξουν το αρχικό κόστος. Ο φίλος μας ε, Βαντελού είπε ότι το φυσικό αέριο και το CCS είναι η λύση για τη μετάβαση από σήμερα σε μια οικονομία με χαμηλό άνθρακα. Συμφωνώ, αλλά δεν θα περιοριστούμε σε αυτά. Θα συμπεριλάβω και την πυρηνική ενέργεια, την οποία δεν ακούσαμε πολλά πράγματα σήμερα και η οποία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ε, παράγει ενέργεια με ελάχιστη ε, δημιουργία διοξίδιο του άνθρακα. Βέβαια τα CCS ε, είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ακόμα πώς δουλεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω να μας αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Τώρα για τη χαμηλή τιμή του άνθρακα και την υψηλή τιμή του πετρελαίου. Εγώ δεν ανησυχώ για την υψηλή τιμή του πετρελαίου γιατί έτσι θα αναζητήσουμε άλλες πηγές ενέργειας. Συμφωνώ μαζί σας και ανησυχώ όμως για τη χαμηλή τιμή του άνθρακα τελικά. Ε, νομίζω ότι ο καθορισμός των τιμών με ρυθμιστικές αρχές είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από μας. Συμφωνώ λοιπόν με τα σχόλια που έγιναν και για το σύστημα ETS. Αν το ETS λειτουργήσει αποτελεσματικά, τότε είναι σαφές ότι θα συμπιέσει την κατανάλωση καυσίμων πλούσιων σε διοξίδιο του άνθρακα. Μου άρεσε ιδιαίτερα και η πρόταση για τη χρήση του διοξιδίου του άνθρακα για να απαγώνουν τα τρόφιμα. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρακτική ιδέα και περιμένω από το κοινό να μας πει εφόσον είναι τόσο κακό γιατί να το χρησιμοποιούμε για να παγώνει τρόφιμα. Να λοιπόν και άλλο ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να καταστήσουμε πιστικό. Ένας άλλος ομιλητής είπε ότι πρέπει να ηγηθούμε αυτή της βιομηχανικής επανάσταση. γιατί αν είμαστε ηγέτες στην αρχή μιας νέας διαδικασίας όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Το θέμα είναι ότι η ιστορία λέει ότι αυτοί οι οποίοι εισέρχονται μετά από τις τεχνολογικές αλλαγές είναι αυτοί που ωφελούνται περισσότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ε, καλή τύχη σε όσους οι οποίοι θέλουν να είναι πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει η υπάρχουσα τεχνολογία. Ο κύριος Όρενσεν είπε ότι απαιτούνται ισχυρότερες κυβερνήσεις για να πετύχουμε τους στόχους μας. συμφωνώ μαζί του. Αγχώνομαι όμως ε, για το τι μπορεί να κάνουν ισχυρές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους χωρίς κυβερνήσεις. Πράγματι ήσασταν αρκετά προκλητικός. Καλό για τη συζήτηση, κυρία Χέρτσοντ, αλλά και κάποιος εκεί στο βάθος, ο 205, έχει ζητήσει το λόγο. Όχι, λάθος. Λοιπόν, η κυρία Χερτσοκ. Ευχαριστώ τους οργανωτές. Είναι πολύ ενδιαφέρον το να είμαστε εδώ σήμερα. Δεν ξέρω αν ήμουν πολύ προκλητική ε, που έθεσα τα ερωτήματά μου ε, νωρίτερα. Εμείς Προχωράμε προς την ευημερία με χαμηλή ε, περιεκτικότητα σε άνθρακα. Όσο καιρό είμαι εδώ και ακόμα και νωρίτερα δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Η καμπύλη των επενδύσεων στον τομέα είναι πολύ χαμηλή και γενικά οι επενδύσεις σε πάρα πολλούς τομείς είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μόνο οι νέες επενδύσεις θα μας οδηγήσουν σε χαμηλότερες ε, εκπομπές. Το θέμα είναι οι επενδύσεις αυτές να οριμάσουν και να αποδώσουν. Εγώ σαν μηχανικός, σαν νοικοκύρα, ξέρω ότι το νερό βράζει στους 100 βαθμούς σαν παράδειγμα, ανάλογα με την εξωτερική πίεση βέβαια. Αλλά η ερώτησή μου είναι αυτή. Πότε πιστεύετε εσείς ε, ε, ότι θα φτάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο και τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Πότε θα έρθει ο βρασμός του δικού μας αυγού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να απενέσω την τόλμη του πρόεδρου μας, του κυρίου Μπούζε, που προχώρησε με την ιδέα αυτής τη διάστασης για την ε, μικρή καταναλωσή άνθρακα και να ενώσει τους τρεις προέδρους και την, ε, τον πρίγκιπα της Ουέλιας ε, με στόχο του με 2050. Έχετε προστάσει σας πολλά μέλη της επιχειρηματική κοινότητας που ήρθαν εδώ, ορισμένοι μας μιλήσαν, υπάρχουν και άλλοι. Δυστυχώς πολλοί από τους συναδέλφους έχουν φύγει, αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε και άλλες αναλογές απόψεων σαν τη σημερινή για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στην οικονομία της, ε, που διέπει αυτή την οικονομία με χαμηλή κατανάλωση ανθρακά για να μπορέσουμε να πούμε περί τίνος πρόκειται και στους νομοθέτες και στον καταναλωτή, αλλά να έχουμε μια ανταλλαγή απόψη με τους ηγέτες της ε, βιομηχανίας μας, ε, να δώσουμε το καλό παράδειγμα μετά. Ξέρουμε ότι λίγες χώρες έχουν δυσκολίες να περάσουν στην ε, οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. θα ρωτήσω τον δόκτωρα Έντιν Χόφερ, για κύριε Πρόεδρε Γιούρσοκ, πώς θα παρουσιάσετε το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι η Πολωνία έχει κάποια προβλήματα. Πώς ε, θα διαμορφωθεί ο δρόμος μέχρι να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουμε και πώς θα τους το εξηγήσουμε καλύτερα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Επνά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές γιατί πιστεύω ότι μεταξύ των παρόντων κανένας δεν θα μείνει δυσαρεστημένος, κανένας δεν θα φύγει δυσαρεστημένος. Το θέμα εξετάστηκε μέσα από διάφορες οπτικές και τρόπους. Εμείς μιλάμε για ε, μια πράσινη οικονομία χωρίς άνθρακα με πράσινη ανάπτυξη τώρα για τις οικονομίες. Η γιαγιά μου έλεγε μη σκέφτεσαι πόσα θα ξοδέψεις αλλά πόσα θα εξοικονομήσεις. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε φαντάζομαι και εγώ με την ενέργεια. Εμείς, ε, άμα δούμε τι ξοδεύουμε, ξοδεύουμε πάρα πολύ ενέργεια στα κτίρια με την αναπαλαίωση, με την θέρμανση, με τις, λαμ... με τις λάμπες, αλλά εγώ ρωτώ, ε, όντας πεπισμένοι εμείς πώς μπορούμε να πείσουμε τους άλλους. Επόμενο σημείο. Πολλοί θύμισαν ότι ο άνθρακας δεν είναι κακό πράγμα αυτό καθεαυτό. Αλλά χρειάζονται καινοτομίες. Και αυτό το οποίο ρώτησε η προλαλή σας ασυνάδελφος είναι πολύ σημαντικό και μέρη απαντήθηκε από τους ομιλητές. Εσείς ε, θυμήσατε ότι οι νόμοι και οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται τάχιστα και με κουράγιο. Χρειάζεται όμως και μία νομοθεσία σταθερή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους διάφορους εδώ στο πάνω και για τον Τζάιλ που πρόκειται. την συζήτηση. Εγώ θα έλεγα να κυριθούμε τώρα αντίστροφα. Ένα λεπτό ο καθένας εδώ για να απαντήσει, για να καλύψουμε το χαμένο καιρό. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τον κύριο Σόρενσον. Ένα λεπτό για να σχολιάσετε αυτά που είπε ο Τζάλ ή οτιδήποτε άλλο αναφέρθηκε από το ακροατήριο. Κύριε Σόρενσον, έχετε το λόγο. όσον αφορά την ανησυχία και την τις κυβερνήσεις που ε, μεγαλώνουν τόσο πολύ που πνίγουν ε, τις πρωτοβουλίες. Εγώ θα έλεγα ότι εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η μόνη αρχή που μπορεί να μας προσφέρει την, το απαραίτητο πλαίσιο, την απαραίτητη δέσμηση που χρειαζόμαστε. 10, 15, 25 χρόνια πολλές φορές ε, χρειάζεται να περάσουν για να λειτουργήσει και αυτό δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει χωρίς κάποιο πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η κυβέρνηση. Αλλά όσον αφορά την νομοθεσία, η ευφυής νομοθεσία είναι αυτή που είναι σημαντική. Χρειαζόμαστε νομοθεσία, οπωσδήποτε. Ευφύη όμως, όπως σας είπα. Πολύ έντονο το μήνυμα αυτό. ο και τη επιτροπή Επιτροπής χρησιμοποιείται όλο αυτό τη υφίους ε, νομοθεσία. Μα ρωτήσετε κατά πόσο ε, το ε, νερό βράζει. Η επιστήμη ναι, το νερό τη κλιματική αλλαγής βράζει. Και αυτό που θέλουμε είναι εκείνοι που είναι και τέστε που προσπαθούν να ρίξουν πάγο στη φωτιά δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Αλλά όταν περνάμε στην, στην οικονομία, πάλι βράζει το νερό. Α δούμε στην Κίνα. 50% τη αιωλική ενέργεια ε, ανά τον κόσμο θα εγκαθιστεί στην Κίνα. Ε, 60-70% τη ενεργή παραγωγή στον κόσμο είναι στην Κίνα είναι η πρώτη χώρα όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η Κίνα. Η Κίνα προωθεί την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας ξεκινώντας από χαμηλά, αλλά προωθεί με μεγαλύτερη επιθετικότητα και αποτελεσματικότητα από ότι οπουδήποτε αλλού. Όσον αφορά λοιπόν την βιομηχανική επανάσταση, βράζει το νερό πράγματι και θα χάσουμε εάν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ναι, ναι, πολύ καλή αυτή η απάντησή σας. Νομίζω ότι το θέμα είναι πώς να περάσουμε και να κάνουμε το όραμα, το όνειρο καλύτερα σε πραγματικότητα, πραγματικότητα. Και εγώ είμαι πεπισμένος ότι έχει επέλθει βλέον το σημείο βρασμού και πρέπει να αντιδράσουμε. Το θέμα είναι αν μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτή τη φάση σωστούς νόμους και μεταβατικές ρυθμίσεις. Σαν παράδειγμα, αν έχει επενδύσει κανείς σε πυρηνική μονάδα, ο χρόνος απόσβεσης είναι 50 χρόνια. Αν θέλει κανείς να δει τι γίνεται μετά από 10 χρόνια θα πρέπει να το κλείσει κανονικά ένα σούπερ μάρκετ είναι 10 χρόνια η απόσβεση της επένδυσης. Πρέπει να, λοιπόν, πάρα πολύ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε την επένδυση στη μεταβατική αυτή περίοδο. Ξέρουμε ακριβώς πόσο περίπλοκα είναι τα θέματα που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ε, από άνθρακα στην Πολωνία, σαν παράδειγμα. Ο περισσότερος κόσμος λοιπόν απαιτεί ότι θα πρέπει στις ρυθμίσεις μας τις νομικές να φανούμε πιο πρακτικοί. Δύο σχόλια. Πρώτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για το συνδυασμό υψηλή τιμή πετρελαίου και χαμηλή τιμή άνθρακα. Η υψηλή τιμή πετρελαίου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους της ανταγωνιστικότητας του άνθρακα και σε παγκόσμια κλίμακα με την Ινδία, τον, τη Βραζιλία, την Κίνα βρισκόμαστε ε, μέσω της αναγέννησης του ρόλου του άνθρακα. Ο μοναδικός τρόπος για να βγούμε από αυτό είναι η σωστή τιμολόγηση του άνθρακα και είμαι πεπισμένος ότι το ευρωπαϊκό σχήμα ανταλλαγής ποσοστώσεων είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Σε άλλο τομέα βέβαια απαιτούνται τρία περαιτέρω βήματα. Το σχήμα αυτό θα πρέπει καταρχάς να συμπεριλάβει και τους 11 τομείς. Όλους τους σχετικούς τομείς λοιπόν. Όταν έχει συμπεριλάβει όλους αυτούς τους τομείς τότε θα έχουμε εγγυήσεις ε, για την υιοθέτηση των ε, τεχνολογιών με λιγότερη χρήση άνθρακα. Θα πρέπει επίσης το σύστημα αυτό να συνδεθεί με τα αναδυόμενα συστήματα ανταλλαγής ποσοστώσεων σε άλλες περιοχές του κόσμου. Θα ήταν εμπνευσμένο θα έλεγα να υπάρξει μια αγορά ΟΣΑ για τον άνθρακα και τρίτον. Η έξυπνη λεγόμενη νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί με σωστό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ρυθμίζουμε όλες τις μεμονωμένες υπάρχουσες τεχνολογίες, αλλά θα έχουμε ένα σχήμα στη διάθεσή μας, τεχνολογικά ουδέτερο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται μια συγκεκριμένη προσπάθεια για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αν εφαρμόσουμε λοιπόν τέτοιου είδους προσπάθειες γρήγορα, τότε θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε από το σημείο βρασμού έγκαιρα και αυτό θα οδηγήσει σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω και τα προηγούμενα πάνελ για τις πολλές πληροφορίες και απαντήσεις που έδωσαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να κάνω δύο μικρά σχόλια. Καταρχάς σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η κυρία Ντίξον Τεκλίβ. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ξέρετε, που ασχολείται με τα θέματα τεχνολογιών και περιβάλλοντος κτλ. Ο πρόεδρος ήταν πριν εδώ άλλωστε. Ασχολείται με τα θέματα αυτά και θα συνεργαστεί μαζί σας. Δεύτερον, νομίζω ότι η αναλογία την οποία έκανε η Χέρτσοκ με το σημείο βρασμού του νερού Νομίζω ότι το θέμα είναι να πείσουμε και τους πολίτες ότι έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση και αυτό δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, πέρα από αυτές τις δύο σκέψεις, λοιπόν, σχόλια, θα δώσω το λόγο για να κλείσει τη συνάντησή μας ο βαριά εργαζόμενος πλέον πρόεδρος μας, ο κύριος Μπούζεκ. Σας ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε αυτού του πάνελ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που μείνανε λίγο παραπάνω, όπως και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην μακρηγορήσω περισσότερο από δύο-τρία λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βασικούς μας ομιλητές και τους επαγγελματίες που ήρθαν εδώ και μας έκαναν τα σχόλια αυτά που ακούσαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που συναντηθήκαμε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Μεταβατική περίοδος για ορισμένε χώρες που βασίζονται στον άνθρακα Λίγες βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς Γι' ε, αυτό είναι απαραίτητο το CCS. Δεν ξέρουμε όμω αν λειτουργεί ή όχι. Να λειτουργεί 100%. Γιατί βέβαια η αποθήκευση είναι το πιο σημαντικό. Γιατί οι τιμέ για τη συλλογή είναι γνωστέ. Ε, το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι τόσο τεράστιο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όμως θα λειτουργήσει γιατί είναι χρήσιμο και για την Κίνα. Και άλλως δεν μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την τεχνολογία. Αδύνατο κάτι τέτοιο. Το δεύτερο θα έπρεπε να είναι βέβαια η ατομική ενέργεια. Όπως είπε ο συνάδελφος Τζάρις Τσίτσεστερ, το κάνουμε στη χώρα μου. ελπίζουμε με μεγάλη επιτυχία. Αλλά θα ήθελα να πω επίση ότι για μικρή περίοδο θα πρέπει να υπάρχει επίσης αποτελεσματική χρήση ενέργειας και εξοικονόμηση. Μπορούμε νομιζω 20, 25, 30, 40% ενέργειας να εξοικονομήσουμε εάν αρχίσουμε σωστή μάχη για κάτι τέτοιο. Τεράστιο δηλαδή. Τεράστιες δυνατότητες. Πάντα το σκέφτομαι αυτό. Και στο τέλος της συζήτησης έχω να πω δύο λόγια μόνο. Ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βέβαια συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, δεν συζητάμε για την επόμενη συζήτηση στη Νότια Αφρική, δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν θα είναι εύκολο, τέλο πάντων. Συζητάμε ένα τέτοιο τεράστιο θέμα για να δούμε πώς θα μπορούμε το θέμα του κλίματος και ε, ε, η, οικονομία με λίγη κατανάλωση άνθρακα. Να το συσχετίσουμε αυτό με την ανάπτυξη, με τη θέση της απασχόλησης και πώς μπορούμε. Καταρχήν να έχουμε μια ενιαία αγορά για την ενέργεια. Αυτό σημαίνει αλληλένδεση. Διαμεθοριακές διασυνδέσεις. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Όχι μόνο λόγω των τιμών, γιατί μια ενιαία αγορά είναι πάντα καλύτερη για τις τιμές. Αλλά επίσης, αυτό ισχύει και για ενιαία αγορά και σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ενιαία αγορά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρει ο συνάδελφος Μαρκολ ε, την έκθεση ότι ενιαία αγορά για την έρευνα και για την ενέργεια, για την ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πράσινη ενέργεια. Μεσόγεια παραδείγματο χάρη, ούτω ώστε η ηλιακή ενέργεια από τη Βόρεια Αφρική να μεταφέρεται στην Ευρώπη ή και ολική ενέργεια από το βορρά της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρώπη με τους διασυνδέσεις αυτές όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και στο ιστορικό κρατών μελών. Και βέβαια να εξαλειφθούν οι νησίδες ενέργειας. Ε, λίγα έχουμε. Οι χώρες γύρω από τη Βαλτική, παραδείγματος, είναι μια τέτοια νησίδα. Και βέβαια είναι σημαντικό αυτό και όσον αφορά τις τιμές, όταν μιλάμε για τους καταναλωτές. Και μετά τους να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Γιατί συζητάμε για την ασφάλεια οδότησης. Και η αγορά είναι σημαντική και από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, οπωσδήποτε πάρα πάρα πολύ σημαντική η ενιαία αγορά. Τεχνολογία, όπως ελέγχθη, να αναπτυχθεί τεχνολογία. Ευρωπαϊκή Στρατηγική ένα πρόγραμμα ορισμένο εγώ είχα πει πριν από τρία χρόνια 10 δισεκατομμύρια θα χρειαστούν γι' αυτό. Φέτο ε, δεν θα φτάνουν. Ε. Edit, 20 θα χρειαζόμασταν. Γιατί έχουμε μια τριών ετών. Χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες, ευρωπαϊκές τεχνολογίες αποτελεσματικότητα. Ατομική ενέργεια, ελληνική ενέργεια, ε, ηλιακή ενέργεια σε 50 χρόνια. Α, σε 50 χρόνια. Καλά. Ας κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή. Και τέλος. Τι θα γίνει με τα χρήματα. Χωρίς τα χρήματα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. 200 δις ευρώ χρειαζόμαστε για τους διασυνθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα θα πρέπει να περάσουν από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά δυστυχώς, ξέρετε, ότι όλα τα σχέδια δεν είναι επαρκώς ελκυστικά για τους ιδιωτικούς επενδυτές. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τα σχέδια αυτά με δημόσιο χρήμα. Λοιπόν, ε, τελική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα πάρα πολύ σημαντικό. Παραδοσιακέ επιδοτήσει χρήσιμο είναι, αλλά θα πρέπει να συνοδεύουν από δημόσια δάνεια και ευφυή χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναπτύξει μια παρόμοια διαδικασία μέσα στα πλαίσια του 7ου προγράμματο πλησίου που λειτουργεί πολύ καλά και οδηγεί σε σημαντική πρόοδο και επενδύσει στον τομέα τη έρευνας και τη ανάπτυξη θα πρέπει να οριστούν στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. και χάρη των νέων τεχνολογιών θα μπορούσαμε να πετύχουμε ανταγωνιστικότητα που είναι πάρα πολύ εύκολο για τους πολίτες γιατί θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε εταιρείε που είναι εδώ γύρω, έχουμε ιδέε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα σωστά νομοθετικά μέσα. Νομίζω ότι συνομιλώντα μεταξύ μα και γνωρίζοντα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ του προβλήματος του κλίματος και του προβλήματος της ενέργειας έχουμε κοινά μία οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα. Γι' αυτό πρότεινα την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας. Πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλιώς θα χάσουμε. Όλα είναι ελεύθερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ, που συζητήσατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεδωθούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ.